So, dear colleagues, welcome back. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε. Μόλις έγινε η ακρόαση μαζί με την Επιτροπή ΑΦΕΤ για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών γενικώ. Και τώρα περνάμε απευθείας στο σημείο 9, συγγνώμη, σημείο 8, την εμπορική πτυχή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα αλλάζω ιδιότητα και θα σας μιλήσω ως ε, εισηγητής. Σας παρουσίασα ένα σχέδιο γνωμοδότησης που βασίζεται και στις δύο πλευρές του νομίσματος η μία πλευρά είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αποτελούν το μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο στις εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις εισαγωγές. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια καλή και σταθερή σχέση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσαν για πάρα πολύ καιρό ε, τον κινητήριο μοχλό εντός του ΠΟΕ. Ήταν και ένας από τους κύριους ιδρυτές ε, του ε, ΠΟΕ και είχαμε και κάποια επιτυχία στις οικονομικές μας σχέσεις. Πολλές συμφωνίες ρυθμιστικής συνεργασίας πέρασαν χάρη στη συνεργασία μας, ε, πιο πρόσφατα μια συμφωνία για, ε, για τον έλεγχο των φαρμάκων ε, στις φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κοινά μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα εμπορίου. Από την άλλη, εμείς διαπιστώνουμε ότι μέσω της νέας κυβέρνησης ε, του κυρίου Τραμπ ε, υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα. Προσπαθεί να υποσκάψει τον ΠΟΕ και θεωρεί ότι είναι η κυρίαρχη αρχή του παγκοσμίου εμπορίου με τους δασμούς ε, για τον χάλιβα και το αλουμίνιο τα οποία επιβάλλει ή το γεγονός ότι δεν δίνει το πράσινο φως ε, για το διορισμό των δικαστών, ε, για το ε, αρμόδιο ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και το όλο σύστημα και επομένως κινδυνεύει στα θεμέλια του το όλο σύστημα. Και επίσης φαίνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν σέβεται τους κανόνες του ΠΟΕ πλέον και προσπαθεί να επιβληθεί μέσω της εξουσίας ε, στην εμπορική πολιτική. Και σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως είναι και λίγο ανησυχητικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται μόνο ε, στα αγαθά, στα εμπορικά αγαθά. Και φυσικά υπάρχουν διάφοροι δασμοί στα αγαθά, αλλά κατά μέσο ώρα οι τελωνιακοί δασμοί είναι λίγο πολύ οι ίδιοι. Κατά μέσο όρο ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε λιγότερο από 1% υψηλότερους δασμούς από ό,τι υπάρχουν στις Πολιτείες. Επομένως, οι διαφορές δεν είναι και πολύ μεγάλες. Ε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες διαφορές βέβαια. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα οχήματα έχει 10%, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 2,5%, αλλά η συνολική εικόνα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν για τα ε, οχήματα τα οποία ε, πολλούνται περισσότερο στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, αυτά τα μικρά φορτηγάκια ένα 25% και επομένω η εικόνα δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Και φυσικά έχουμε και εμπορικές σχέσεις και για τις υπηρεσίες. Οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι μεγάλος προμηθευτής υπηρεσιών και έχουν πολλά χρήματα από ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως υπάρχει μια ευρύτερη εικόνα Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ αυτή τη στιγμή εξετάζει μόνο την εμπορία ε, αγαθών. Πρέπει λοιπόν τελικά να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να αποκαταστήσουμε τη συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Βέβαια θα χρειαστούν πολλές συνομιλίες με τους ενδιαφερομένους στις Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κενό εμπορικό θεματολόγιο για το διμερές εμπόριό μας, αλλά και για να υπάρξει σταθεροποίηση του παγκοσμίου εμπορίου. Και βεβαίως όπου χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε και με τις Ηνωμένε Πολιτείε τι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συζητηθούν καταρχάς και βεβαίω θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και κάποια διμερεί θέματα εμπορίου και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τις τρίτες χώρες σε θέματα διανοητικών δικαιωμάτων ή όσον αφορά την ε, ε, υπερπληθώρα προσφοράς ε, χάλιβα. Αλλά, και αυτό το λέω και στη γνωμοδότησή μου, θέλουμε να υπάρχει εταιρική σχέση. Και δεν θα διαπραγματευτούμε συμφωνία υποπίεση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι οι δασμοί στο χάλιβα και το αλουμίνιο δεν συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ και δεν θα τους δεχτούμε. Πράγματι λοιπόν πρόκειται για ένα νόμισμα με δύο όψεις και πρέπει να επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή στην πιο προβληματική όψη. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στους κοιόδης συζητητές από το ΕΛΚ καταρχάς. απουσιάζει η ε, σκιώδη συγγήτρια, θα μιλήσει ο κύριος Πάμπηξ στη θέση τη. Ευχαριστώ. Έχετε του χαιρετισμού τη Γκοντελίβε Κουίσχα ε, Ρόβολ και με χαρά θα σας διαβάσω τα σχόλια που έστειλε για την Επιτροπή μας. Πρώτον, ευχαριστίες για την προσωπική σας δέσμευση για τα θέματα των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ηνωμένων από την άποψη του ΕΛΚ εμείς λέμε ότι θα πρέπει να είναι ισόρροπη η γνωμοδότηση και πάντα να είμαστε πρόθυμοι να έχουμε σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως θα πρέπει να κοιτάξουμε τις τελευταίες εξελίξεις και να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε στο μυαλό μας ε, το μακροχρόνιο διάστημα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι και θα παραμείνουν σημαντικότατος εταίρος και στο εμπόριο και αλλού. Και δεν χρειάζεται να πούμε ότι ιδιαίτερα στον ΠΟΕ χρειάζεται ισχυρή δέσμευση ε, των ΗΠΑ για να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Θα πρέπει λοιπόν να ε, εξαλείψουμε, να απαλύνουμε αυτές τις εντάσεις που βλέπουμε τώρα στο χάλιβα και το αλουμίνιο για να έχουμε βαθύτερη και στενότερη εμπορική συνεργασία με τους Αμερικανούς μας συμμάχους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Μακλάρκιν από το ECR. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για το σχέδιο γνωμοδότησης. Η ομάδα μας συμφωνεί με τις προτάσεις σας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το ε, αδιέξοδο με τον ΠΟΕ και να διερευνήσουμε και άλλους δρόμους για να ε, προωθήσουμε τις διμερείς μας ε, σχέσεις. Η ομάδα μου ανέκαθεν ήταν αναφανδόν υπέρ των σχέσεων με τις ΗΠΑ και των διατλατικών σχέσεων γενικότερα και μόνο ο όγκος των συναλλαγών που έχουμε, οι δύο πλευρές ε, δείχνουν ότι κάποια συμφωνία χρειάζεται, είτε αυτή είναι η TTIP είτε κάποια άλλη. Βλέπουμε τις πρόσφατες εμπορικές εξελίξεις παγκοσμίω. Και ιδιαίτερα το γεγονό ότι έχουν μπλοκάρει το διορισμό στο πάνελ διαιτησίας ε, του ΠΟΕ. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για όλα αυτά τα θέματα, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και την ευκαιρία αυτή να δούμε πού έχουμε κοινή προσέγγιση και πού μπορούμε να τα βρούμε και να επιτύχουμε κάποια πρόοδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαπραγματευόμαστε ε, με την απειλή όπλου, αλλά πώς ε, θα βοηθήσουμε την οικονομία μας να δούμε και το παγκόσμιο εμπόριο. Υπάρχουν και άλλα μέτρα, μη δασμολογικά, επενδύσεις, δημόσιες συμβάσεις, ε, ψηφιακή οικονομία, ε, διανοητική ιδιοκτησία, για να αναφέρω μερικά και μόνο. Στη γνωμοδότηση θα πρέπει να δούμε και τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί πάντα επικεντρωνόμαστε στους μεγάλους ομίλους και τις επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε ε, μόνο τα εμπόδια που έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην Αμερική, αλλά και το αντίστροφο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. και στι ροές των δεδομένων. Τα ξέρω τα προβλήματα με το χάλιβα και το αλουμίνιο, αλλά ακούμε και διαφορετικές και διάφορες εξελίξεις για ποσοστώσεις που συμφωνούνται κτλ. Βεβαίως υπάρχει υπερβολική παραγωγή χάλιβα να δούμε πώς μπορούμε στο διεθνές πλαίσιο να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε κλιμάκωση του προβλήματος, να παραμείνει ανοιχτός ο διάλογος και βεβαίως το θέμα του ΠΟΕ και αυτή η διάνεξη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το καλύπτει η γνωμοδότησή σας διεξοδικά. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση από κοινού. Χωρί τι ΗΠΑ αποκλείεται να βρεθεί λύση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Βλέπω ότι επιτέλους έχουν διορίσει και πρέσβη στον ΠΟΕ και με χαρά να συνεργαστούμε μαζί του. Ελπίζουμε να δώσουμε πιο θετικό τόνο στη γνωμοδότηση, με τις τροπολογίες, να μιλάμε μόνο τα αρνητικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σχάκε από τους φιλελευθέρους. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ. Πολλά υπόθηκαν. It ε, Μας δίνει την ευκαιρία όμως η γνωμοδότηση αυτή να εκφραστούμε και εμείς ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο για κάποια κομβικά ζητήματα. Ε, όλα αυτά τα δασμολογικά, τα θέματα των κανόνων, η σύγκρουση με τις ΗΠΑ που ζούμε αυτόν τον καιρό θα πρέπει να αναφερθεί. Συμφωνώ με την ΕΜΑ, έχουμε την ευκαιρία να πούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες ε, θα προχωρούσαμε σε διαπραγματεύσεις. Ξέρω ότι οποιασδήποτε συνομιλίες τύπου TTIP είναι τώρα στο ψυγείο, στη, βαθιά κατάψυξη αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε για το πώς, το πότε και να πούμε τη γνώμη μας. Επίσης υπάρχει και το θέμα της ετεροδικίας με τις κυρώσεις. Αυτό επανέρχεται ε, πάντα στη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πούμε ε, πόσο σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενωμένη. Διότι η χώρα ε, που γνωρίζετε καλύτερα η πατρίδα σας ε, κάπως τριμώχνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό δεν βοηθάει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ενωμένη, όχι ο καθένας να προσπαθεί να παίξει το δικό του παιχνίδι. Είναι μια καλή βάση λοιπόν για τη συζήτηση και τη συνεργασία και νομίζω ε, ότι θα στείλουμε μια καλή και ισχυρή γνωμοδότηση στην έκθεση ε, της Επιτροπής Εξωτερικών ε, χωρίς να μαστεγώνουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά να πούμε για τις αρχές, τις αξίες τις οποίες μοιραζόμαστε. Και είναι πολλοί Αμερικανοί ε, οι οποίοι συμφωνούν μαζί μας, άσχετα αν δεν κατοικούν στο Λευκό Οίκο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Ο, ο Γιάννικ Ζαντό που ε, Χέλμουτ Σόλτς, την Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλις ε, ερχόμαστε από την κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Εξωτερικών και βλέπουμε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το θέμα των διατλαντικών σχέσεων και έχω λίγο την εντύπωση ότι δεν έχουμε συζητήσει ακόμα σωστά το μέγεθος ε, και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ε, σωστή είναι η γνωμοδότησή σου για την Επιτροπή Ίντα, συμφωνούμε ιδιαίτερα με το σημείο 1, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι αν δεν ήταν τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά μια άλλη χώρα με την οποία θα συζητούσαμε, που θα ήταν η πιο αδύναμη, θα είχαμε ε, τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Από ό,τι φαίνεται όχι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η παριθμόν ένα εξαγωγική αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερη εισαγωγική, δηλαδή εξάγουν σε εμά. Αυτά είναι κάποια οικονομικά δεδομένα και πραγματικότητες που αφορούν επιχειρήσεις μεγάλες, μεσαίες και μικρές. Και μεγάλη πρόκληση για τις εταιρείες αυτές και, και για μας, τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε, σωστό είναι να διατρανώσουμε με την γνωμοδότηση ότι θέλουμε ένα εμπορικό σύστημα που να βασίζεται σε κανόνες και να διέπει ε, υποχρεωτικά και τις σχέσεις ε, Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να διατηρήσουμε στη ζωή, το λέω έτσι προσεκτικά, αυτό το σύστημα του πολυμερούς εμπορίου. Ενδιαφέρον βρίσκω το γεγονός ότι η γνωμοδότηση ασχολείται και με το γεγονός ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο το πάνελ διατησίας του ΠΟΕ, ακόμα και απουσία των Ηνωμένων Θα πρέπει να σταθεροποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας και να εξασφαλιστεί του ΠΟΕ. Κάτι άλλο που θα έλεγα ακόμα ε, και είναι σημαντικό για τη συνεργασία μας και για τις εργασίες μας εδώ δεν θα πρέπει να συζητάμε μόνο με τις Ηνωμένε Πολιτείε για τη μεταξέλιξη του πολυμερού εμπορικού συστήματος, αλλά και με άλλους συνομιλητές και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και να ασχοληθούμε με τις εξελίξεις, διότι μόνο έτσι θα λυθεί αυτό το θέμα από κοινού με όλα τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ για να έχουμε ένα πολυμερές σύστημα εμπορίου, να διατηρηθούν οι δομές, όχι για το εμπόριο το ίδιο, αλλά γιατί έχουμε και παγκόσμιες προκλήσεις. Αυτό μου λείπει από την γνωμοδότηση, μάλλον μου λείπει από την ε, στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια θα έχουμε σχέσεις και θα συζητήσουμε τα κριτήρια για την εμπορική και οικονομική γενικότερη συνεργασία. E Τιτσιάνα για το e Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, επεσήμαναν πολλοί συνάδελφοι, οι σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, βρίσκονται σε μια κατάσταση που ποτέ ήταν τόσο ανησυχητική. Και πέραν το γεγονό ότι πλήττεται η παραγωγή μα ε, χάλευα και αλουμινίου, απειλούν και την αυτοκινητοβιομηχανία και την αγορά φαρμάκων και τελευταία υπόθεση Airbus ε, που έκλεισε χθε από τον ΠΟΕ, η οποία επιδεινώνει περαιτέρω την ευρωπαϊκή θέση. Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει και τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει που έχουν ε, εμπορικέ σχέσει με το Ιράν. Και φυσικά αυτό πλήττει κυρίω κάποιε χώρε όπω είναι η Γερμανία και η δική μου ε, είναι σαφές λοιπόν ότι η αμερικανική ε, στρατηγική είναι να κατακαιρματίσει το ευρωπαϊκό μέτωπο, να βάλει τη μία χώρα εναντίον της άλλης και ε, να υπάρξει και μια εμπορική αντεπίθεση. Είπατε πολύ καλά πώς έχει κατάσταση και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό ε, με αυτά που είπατε. Πρέπει να επαναφέρουμε το ρόλο του ΠΟΕ αυτή τη στιγμή, να φροντίσουμε να συμμορφωθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε στους ελάχιστους κανόνες που υπάρχουν για το διεθνές εμπόριο και να μην υπάρχουν μονομερείς δράσεις. Αν και αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρει ο ΠΟΕ να αντιδράσει εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης την σημασία να παραμείνει ενωμένη η Ευρώπη και να μην σκύψει το κεφάλι σε αυτά τα αιτήματα, γιατί θα ανοίξουμε την ε, πόρτα για περαιτέρω απαιτήσει στο μέλλον. Φαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση η Ευρώπη είναι μια χώρα σαν όλες τις άλλες και όχι ένας προνομιακός εταίρος. Ίσως ε, φταίει και η Ευρώπη η οποία δεν μπορεί να ακολουθήσει μια κοινή γραμμή. Αλλά πιστεύω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να καταλάβουν ότι θα είμαστε πιστό του σύμμαχο, αλλά πρέπει να είναι και αυτή η πιστή μα σύμμαχοι. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ και τώρα ο λόγο του Βιάννα Ρέντινγκ. Σα ευχαριστώ για όλα όσα έχετε πει ως τώρα. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται κάποια βελτίωση τη κατάσταση, αλλά με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό και πώ θα το πετύχουμε. Σίγουρα όχι με κράτη-μέλη που λειτουργούν μονομερός για να εξάγουν ωφέλη. Μόνο σαν σύνολο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και όχι με διαπραγματεύσει υποποίηση, γιατί τότε μόνο θα, μόνο θα να χάσουμε έχουμε. Πρέπει να είμαστε δυνατοί. Θα πρέπει να έχουμε μέτρα που θα απαντήσουν στα μέτρα τους. Είναι κάτι πολύ σκληρό, αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά αν δεν είμαστε σκληροί θα μας δουν ως αδύναμους, δυστυχώς, και θεωρώ γι' αυτό ότι μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ενισχυθεί ο διάλογος στο Κογκορέσο και αυτό είναι αυτό που θέλουμε όλοι μέσα σε αυτό το χώρο για να βελτιώσουμε τις σχέσεις πρέπει να πράξουμε το έργο για το οποίο έχουμε εκλεχθεί και θα πρέπει σε αυτό το επίπεδο να παρέμβουμε. Πρέπει όμως να ασκήσουμε και κριτική όταν κράτη-μέλη κάνουν την Ευρώπη πιο αδύναμη με τον τρόπο που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ε, την κατάσταση και να εξάγουν ωφέλη. Μόνο όσο ενιαία Ευρώπη μπορούμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. εκτός μικροφώνου. Είναι, ε, υπάρχει μια σύγχυση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω, ο κύριος Πάμπριξ δεν είναι εδώ, αλλά θέλω να τον συγχαρώ για την πολύ όριμη παρέμβαση του στην ακρόαση προηγουμένως Έχουμε όλοι των πρώτων των ΗΠΑ, αλλά θα ήθελα να πω το εξή. Δεν μπορούμε πάντα να είμαστε αρχηγό τη χώρα μα. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε το δικό μα αρχηγό χώρα. Πώ να επιλέξουμε τον αρχηγό μια άλλη χώρα. Άρα όποια κριτική και να ασκήσουμε δεν έχει σημασία. ως μέλος του Independence Party δεν θα έχω ποτέ έναν αρχηγοκράτη που τον εγκρίνω. Να συγχαρώ τον Πρόεδρο για την γνωμοδότηση που είναι πλήρης και μελετημένη. Το γενικό πλαίσιο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει ένα έλλειμμα 147 εκατομμυρίων και 55 εκατομμύρια πλώνασμα στις υπηρεσίες. Δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κυμαίνεται ο διάλογος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου αρέσουν οι Financial Times, αν και διαφωνώ με όλα αυτά που πρεσβεύουν. Υπάρχει ένας γερμανός σχολιαστής της ε, Financial Times, ο οποίος ε, ε, δημοσίευτα αυτό τη Δευτέρα. Αναφέρει συνεχώς, επανειλημμένος, με πολύ μεγάλη σαφήνεια και βασιζόμενος σε γεγονότα ότι η Γερμανία έχει πλεονάσματα στις εξαγωγές αγαθών, υπερβολικό πλεόνασμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την υγεία της οικονομίας και για την ευημερία της γερμανικής οικονομίας και τους ε, ανθρώπους που ζουν εκεί. Είμαι υπέρ της Γερμανίας, φίλο Γερμανός, Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη συζήτηση. Και θα ζητήσω από τον πρόεδρό μας αυτά τα βασικά γεγονότα να εκτεθούν, να γίνει αναφορά σε αυτά γιατί κατά τα άλλα είναι μια πλήρης και πολύ καλά βελτιμένη γνωμοδότηση. Κύριος Μογέλα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν σε αυτή την έκθεση μπορούμε να βάλουμε στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της Γερμανίας. Μπορεί να το, στείλουμε, να το παραπέμψουμε σε άλλη συζήτηση. Συμφωνούμε βεβαίως με τη γνωμοδότηση. Είναι σωστή η διάγνωση και για την πραγματικότητα των διατλαντικών σχέσεων που είναι έντονες και σημαντικές αλλά ταυτόχρονα και ε, ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κανείς δεν αμφισβητεί την εκλογή του κυρίου Τραμπ αλλά ε, ε, με την έλευσή του στην εξουσία στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ήρθαν και τα μεγάλα προβλήματα. Ο ΠΟΕ, οι δασμοί, δεν δίνει ε, το πράσινο φως για το διορισμό δικαστών στα διαιτητικά όργανα. Και ε, κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ, πολύ ωραία το είπατε, θέλει να κάνει επίδειξη δυνάμεως. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, έχουμε τώρα την ευκαιρία να δείξουμε ότι θα δοκιμαστεί η, η εξουσία μας και η δύναμή μας, αλλά θα αντέξει ούτε τι πλάι θέλουμε, ούτε συμφωνία για τις ποσοστώσεις, ας πούμε, για να ε, μειωθούν οι ε, δασμοί για το χάλιβα. Θα πρέπει να είμαστε στεναροί, να μην ε, γονατίσουμε και να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στην ισχύ και στη δύναμη της Ευρώπης. Το είπε θαυμάσια η κυρία Ρέντινγκ. Το πρώτο που θα πρέπει να αποφύγουμε είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε να αρχίσουν διμερείς επισκέψεις να επιδίδονται σε αυτές, αλλά να είμαστε ενωμένοι και στοιχημένοι. Και υπάρχει μια ελπίδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει εδώ. Και μπορεί να είναι το τέλος της θητείας, μπορεί το Κοινοβούλιο να έχει ως θεσμικό όργανο τα όρια του, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα όλες οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να διατρανώσουμε ξανά αυτή την ισχύ της Ευρώπης. Αλλιώς η διαπραγμάτευση θα είναι τελείως ετεροβαρής και θα χάσουμε κατά κράτος. Ευχαριστώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωστός και μη εξαιρεταίος Κίντο Χούμπερ από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε σχόλια για την, γνωμοδότησή σας προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυτό είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο νέο για μένα. Είναι καλά νέα. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τα σχόλια. Είχα περιορισμού στον ετοίμασα αυτή τη γνωμοδότηση ένας περιορισμός ήταν ε, περιορισμένος χώρος και το δεύτερο ήταν ε, ο χρόνος. Γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι αυτά που γράφει είναι πάντα σχετικά ε, για επικαιρά την επόμενη μέρα. Όσον αφορά το θέμα της ενότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήμουν πολύ ε, κατά τη σύνταξη γιατί υπήρξε ενότητα. Προσπαθώ πάντα έναν τρόπο για να αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες και φυσικά πρέπει να εμείνουμε στην ενότητα και την ξεκάθαρη προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι σχετικό για σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω και για τα υπόλοιπα ερωτήματα που τέθηκαν για την εξωτερικότητα και τον δίκτυο που μπορεί να έχουν κάποια μέτρα των ΗΠΑ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επίσης όσον αφορά τις μελλοντικέ σχέσεις Και επίση το έρωτο που κάνετε για τα αντίπεινα μέτρα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε στην γνωμοδότηση και είμαι πρόθυμος και έτοιμος να δω τις ε, προτάσεις τροπολογίας σας και είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε μια ισχυρή φωνή, θα βρούμε ε, συμβαστικές προτάσεις Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 26 Μαΐου στις 6 ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο σημείο 9 της μερίσιας διάταξης. Αξιοποιώντας την παγκοσμιοποίηση, εμπορικές πτυχές, είχαμε μια ανακοίνωση στην Επιτροπή και κάποια νέα στοιχεία ε, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση. Ο εισηγητής μας είναι ο Γιώαχιμ Σούστερ. Του δίνω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Μπεάντ. Θεωρώ ότι το έγγραφο προβληματισμού δεν ήταν ξεκάθαρο ως προς ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε ήταν άλλη του 2017, στο μεταξύ εξελέγει ο Τραμπ, αλλά δεν ήταν ποτέ ξεκάθαρο τι θα συμβεί όσον αφορά το εμπόριο. Κάνουμε πάλι λόγο για εμπορικούς πολέμους και θεωρώ ότι, ότι αυτό που τελευταία ισχύει σε καμία περίπτωση ο κύριος Τραμπ δεν ε, μπορεί να περιοριστεί και ούτε ο κόσμος θα γίνει καλύτερος άμα δεν επανεκλεγεί. Όλα αυτά αφορά το έγγραφο προβληματισμού εμπόριο και παγκοσμιοποίηση. Είναι εξαιρετική η παρουσίαση του και μας ε, ε παροτρύνει να δημιουργήσουμε μια καινούργια στρατηγική. Από τη δικιά μου οπτική και την παρουσιάζω και στην έκθεση υπάρχουν τρεις βασικές προκλήσεις οι οποίες έχουν συνεπίσει είναι τα προτερήματα της ε, παγκοσμιοποίησης για τον πληθυσμό και μεταξύ περιφερειών υπάρχει άνηση, άνησος καταμερισμός. Υπάρχει αυτή η ανισότητα που έχει οδηγήσει και σε πολιτικές αντιδράσεις σε πολλούς ε, τομείς. Ένα σημείο ε, είναι το θέμα του Τραμπ το δεύτερο. Έχει να κάνει με ε, τη μετατόπιση του κέντρου βάρους ε, την ε, άνοδο της σημασίας των ε, ασιατικών χωρών και κυρίως της Κίνας ε, γιατί κερδίζουν έδαφος και στην οικονομία και στην πολιτική και ποια είναι η σχετική απώλεια που θα έχει η Ευρωπή και η Βόρειος, Βόρεια Αμερική και ταυτόχρονα και είναι το τρίτο σημείο είναι η παγκόσμια οικονομία και η παγκόσμια οικονομική τάξη όπως ε, σχηματίστηκε με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πώς απεικονίζονται τα συμφέροντα των διάφορων ε, κρατών. Υπάρχει ένας απορτουνισμός. Θα πρέπει λοιπόν Και σύμφωνα με αυτές τις τρεις ε, τάσεις θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, όπως παρουσιάζεται στο έγγραφο προβληματισμού, να αναπτύξουμε μια απάντηση σε όλα αυτά. Είναι απαραίτητο πάντα το έγγραφο αυτό για το εμπόριο είναι αρχή του 2015. Θα πρέπει λοιπόν να ε, λάβουμε υπόψη ε, σε αυτό το έγγραφο και τους ε, στόχους της ε, στόχους βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια στρατηγική απάντηση στις νέες προκλήσεις κατά πρώτον να ενσχυθούμε εσωτερικά αυτό πρέπει να το αντικατοπτήσουμε και στην έκθεση, στη δικιά μας εσωτερική αγορά, την νομισματική ένωση, αλλά και ταυτόχρονα να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε ε, παγκόσμιο επίπεδο ε, και στην ψηφιοποίηση, να ανανεώσουμε την ε, ενεργική μας βάση και αυτό με προστατευτικά μέτρα, τα οποία επίσης τα χρειαζόμαστε, μέτρα προστασίας του εμπορίου θα μιλήσουμε και για το greening στις επενδύσεις. Όμως είναι απαραίτητο να έχουμε διαδεθοντικά μέτρα προσαρμογής και να λάβουμε υπόψη σε αυτά και τις ε, ε, περιφέρειες οι οποίες αδικούνται. Πρέπει να τονίσουμε την πολυμερή, τον πολυμερή χαρακτήρα των αντιπραγματεύσεων, αλλά να είμαστε και αρκετά μαχητικοί σε περίπτωση διμερών διπραγματεύσεων. για να επιδιώξουμε και να συνδέσουμε και τους ε, στόχους της βιωσιμότητας και να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο να λάβουμε ισχυρά υπόψη τους, τις τονικές χώρες μια προοπτική ανάπτυξη στο εμπόριο με τις αφρικανικές χώρες. Θεωρώ όμως ότι είναι επίσης λογικό να ε, ενισχύσουμε και την πολιτική προς την ε, Ανατολή και να συμπεριλάβουμε μια προσπάθεια για μια ε, πιο ισχυρή συνεργασία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια στρατηγική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. Αυτά συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο προβληματισμού. και μπορούμε να πούμε ότι από τη μια πλευρά ε, έχει μια πολύ καλή προσέγγιση το έγγραφο αυτό, αλλά υπάρχουν ε, και κάποια άλλα σημεία στα οποία θα πρέπει να τονίσουμε συγκεκριμένους τομείς και να επεκταθούμε. Αλλά χαίρομαι ε, πάρα πολύ ε, για έναν ενδεχόμενο διάλογο, για στρατηγικό διάλογο, ώστε να προσδιορίσουμε τα αδύναμα σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα σκιώδη συζητητές. Κυρία Νεκμίνε για το EPP. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν κίνδυνοι κατά της παγκοσμιοποίησης, οι συμφωνίες ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά οδήγησαν σε διαδηλώσεις και αυτό φυσικά ε, οδήγησε και σε σταδιακές αλλαγές ε, στον τόνο μας. Το έγγραφο προβληματισμού του Μαΐου του 2017 για την παγκοσμιοποίηση δείχνει πώς θα μπορούσαμε ίσως να απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις και ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να αναγνωρίσει ε, και το αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Πρέπει λοιπόν τα ωφέλη της παγκοσμιοποίησης ε, να ε, κατανεμηθούν πιο δίκαια. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα σε απάντηση στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή των κανόνων για να μην ε, υπάρχει κίνδυνος μείωσης των μισθών, ε, επισφαλή συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους, ε, dumping και εκμετάλλευση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σταματήσουν τις άδικες πρακτικές και οι πολυεθνικές θα πρέπει να είναι υπόλογες πλέον για την φοροαποφυγή και την παράκαψη του εργατικού δικαίου. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όταν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιχειρούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους ε, μέσω της αλυσίδας διανομής. Πρέπει να καθησυχάσουμε τους πολίτες μας ότι η χάραξη πολιτικής έχει κάποια πλέον μέτρα ε, και οι θύνοντες έχουν μέτρα στη διάθεσή τους για να προχωρήσουν σε κάποια πράγματα. Και το εμπόριο είναι απλώς μια πτυχή ενός ευρύτερου φαινομένου της παγκοσμιοποίησης. Τα ε, πλήθη τα οποία συγκεντρώνονται σε, όλη την σε όλο τον κόσμο οι Αυστραλοί που βλέπουν το διαγωνισμό της Eurovision στη Λισαβόνα, όλα αυτά είναι παγκοσμιοποίηση. Και ο διασυνδεδεμένος κόσμος μας. Οι τεχνολογίες προσεγγίζουν τους ανθρώπους, η οικονομία και η αλυσίδα διανομής αλλάζουν επίσης, η αλυσίδα προμηθειών, συγγνώμη, και φυσικά προχωρούν πολλά πράγματα σε πολλές χώρες. Στον κατασκευαστικό τομέα θα μπορούσε αυτό να είναι απειλή λόγω της αυτοματοποίησης, αλλά ο προστατευτισμός είναι Μία απάντηση η οποία δεν ε, είναι κατάλληλη για την παγκοσμιοποίηση. Το να κλείσουμε τα σύνορα και να έχουμε παγκοσμιοποίηση θα οδηγήσει σε φαινόμενο ντόμινο για όλου, θα ζημιώσει του εισαγωγεί, του εξαγωγεί και του καταναλωτέ. Επομένω, οι εμπορικέ μα συμφωνίε βοηθούν ε, ε, τι επιχειρήσει μα να παραμείνουν ανταγωνιστικέ ανά τον κόσμο. Αλλά έτσι συμβάλλουμε και στη διαμόρφωση τη παγκοσμιοποίηση προ το καλύτερο. Οι εμπορικέ μα συμφωνίε περιλαμβάνουν δεσμεύσει και για τι δύο πλευρέ, μέσω των υψηλότερων περιβαλλοντικών στόχων και προτύπων υγείας. Και πρεμένως έτσι μπορούμε να εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και ε, να υποχρεώσουμε τις ξένες κυβερνήσεις να σταματήσουν τις φθηνές εξαγωγές προς την Ευρώπη. Και επομένως πρέπει να βρούμε μια απάντηση για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης, ε, δεδομένου ότι το 1 τρίτο του εισοδήματος των κρατών μελών προέρχεται από εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο. Η ε, αντιμετώπιση λοιπόν της παγκοσμιοποίησης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το διεθνές εμπόριο, αλλά δεν θα πρέπει να φοβούμαστε την παγκοσμιοποίηση, γιατί όλα τα εργαλεία τα έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει απλώς να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και εμείς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμφωνήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι πρέπει να δράσουμε κατεπηγόντως και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε από κοινού. Εκ μέρους του ΕΛΚ, λοιπόν, προσβλέπω στη συνεργασία μας ε, για το θέμα αυτό. Τέλεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα μας καλωσορίζει το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διθάσευση της παγκοσμιοποίησης και συμφωνούμε με πολλά στοιχεία και με τους στόχους. Είναι σαφές ότι η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος δημιούργησαν ε, πολλές ευκαιρίες για καταναλωτές και για επιχειρήσεις. Και τώρα είναι παγκόσμιο το εμπόριο και ε, τα καταναλωτικά αγαθά ε, μπορούν να αγοράζονται, να πολλούνται παγκοσμίω. Τα δεδομένα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Οι καταναλωτές θέλουν όλο και νέα προϊόντα. Έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση και δημιουργήθηκαν τεράστιες ευκαιρίες. Αλλά με τις ευκαιρίες έρχονται και οι προκλήσεις και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είμαστε σε θέση να τις αντιμετωπίσουμε. Όπως είπε και η συνάδελφος, υπάρχει και η άλλη πρόκληση της κοινή γνώμης. Και όλο και περισσότερο ο κόσμος κατηγορεί το εμπόριο για προβλήματα ε, στο εργατικό δίκαιο, για τις απώλειες θέσεις απασχόλησης, ε, και γενικά για την οικονομική του κατάσταση. Πρέπει να τους πείσουμε ότι είναι καλό το εμπόριο και δεν φταίει το εμπόριο. Να υπάρχουν μηχανισμοί προστασίας του εμπορίου όσο γίνεται διαφανέστερες διαπραγματεύσεις, ε, βελτίωση ε, των διαδικασιών, μείωση των εμποδίων των κανονιστικών και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται στραμμένη προ τι νέε τεχνολογικές εξελίξεις και το ψηφιακό εμπόριο. Όσο και αν σκεφτόμαστε και τα περιβαλλοντικά θέματα και τα κοινωνικά και τη βιωσιμότητα. Ελπίζω ε, οι προτάσει μας να βρουν χώρο στο σχέδιο της έκθεση. Ευχαριστώ από του πράσινου, η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Το έγγραφο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θάσευση της παγκοσμιοποίησης σε εμπορικές πτυχές είναι μια πολύ καλή ε, συμπλήρωση ε, ε, του σχεδίου που έχει για το εμπόριο για όλους. Ωραίες είναι αυτές οι ιδέες, αξιέπαινες και αξιόλογες, αλλά πώς θα κάνουμε τον κόσμο να τα αποδεχτεί. Uh, και πώς ε, μπορεί ο πλανήτης μας να γίνει πιο βιώσιμος. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι τι ρόλο έχει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομοθέτης. Δηλαδή να, καθορίζει εκείνη το παιχνίδι και τους κανόνες και όχι να υφίσταται αποφάσεις άλλων. Δύο παραδείγματα ίσως. Ο κανονισμός, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων αυτή τη στιγμή είναι ένα παράδειγμα ότι η Ευρώπη θα καθορίζει παγκοσμίω ε, τους κανόνες και τις νομοθεσίες και πρέπει να το έχουμε υπόψη. Έχουμε το δυναμικό αυτό, απλώς είναι αναξιοποιητό, δεν το εκμεταλλευόμαστε πλήρως. Άλλο παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια είναι πρωτοπόρα σε ε, θέματα κλίματος και πολιτικές και χάρη σε εκείνη γεννήθηκε και η Συμφωνία των Παρισίων με τη μορφή που έχει. Και θα πρέπει όλα αυτά τα επιτεύγματα να ε, βρίσκουν το χώρο που τους αναλογεί ε, και να αντανακλώνται και στις εμπορικές πολιτικές. Ποιο είναι το ερώτημα λοιπόν, πώς μπορεί και πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει αποτελέσματα στις ιδέες που προτείνει στο έγγραφο αυτό. Παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία τα έχετε σε πρώτη γραμμή. Στην πράξη τι κάνετε, γιατί δεν έχουμε δει και πολύ μεγάλες αλλαγές. Ε, ε, και έχουμε και κεφάλαια για βιώσιμη ανάπτυξη ε, στις εμπορικές συμφωνίες, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει λήξει η συζήτηση για την επιβολή κυρώσεων και για την υλοποίηση αυτών των συμφωνιών και από τις τρίτες χώρες. Σήμερα το πρωί είχαμε μια πολύ καλή ε, συζήτηση σχετικά όταν συζητούσαμε τον εξχρονισμό της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού, που νομίζω ότι είναι μάλλον φρούδα, ελπίδα και κενή υπόσχεση για τα θέματα αυτά της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάποιο βαθμό ενδεχομένω τους πρασίνους έχει γίνει ένα μεγάλο καινοτόμο βήμα έτσι ώστε ε, τα κοινωνικά θέματα, τα περιβαλλοντικά θέματα και η καταπολέμηση του ντάμπινγκ και τα σχετικά ε, μέσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτής της μεθοδολογίας πώς προτίθεται να τις μεταξελίξει και σε τι χρονικό ορίζοντα. Ευχαριστώ. Και πάλι ο Χέλμουτ Σόλτς από την Ενωτική Αριστερά. Ναι, αλλά θα επιθυμούσα να μιλήσει πρώτα η Αν Μαρή Μαγιόρ και μετά εγώ. Μινέρ, συγγνώμη. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην παρούσα έκθεση δεν επενεί μόνο ε, τα θετικά, ε, αναφέρει και τα αρνητικά. Δυστυχώς όμως τα υποτιμά και δεν ψάχνει λύσεις. Ευνοούνται οι πολυεθνικές και την πληρώνουν οι άνθρωποι, τα ζώα και το περιβάλλον και η δημοκρατία υπονομεύεται, καταργείται, καταστρέφεται η αλληλεγγύη και χάνουμε και τη ε, φύση και το περιβάλλον. Ε, οι διαπραγματεύσεις γίνονται και κλεισμένων των θυρών και διαφεύγουν των εθνικών ε, κοινοβουλίων. Και υπονομεύεται η δημοκρατία γιατί η πολυεθνικές έχουν τον πρώτο λόγο πριν από τους εθνικούς αντιπροσώπους και οι, οι αλλοδαποί ε, επενδυτές έχουν ε, ένα ξεχωριστό σύστημα διατησίας, ένα ξεχωριστό σύστημα επιβολής δικαιοσύνης, στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση ΜΚΟ και άλλοι. Και ποια είναι τα θύματα ή ε, το περιβάλλον. Οι στόχοι της βιωσιμότητας αναφέρονται μεν, αλλά δεν είναι δεσμευτικοί. Οπότε είναι μάλλον διακοσμητικά όλα αυτά. Πρόεδρε, θα πρέπει να ασχοληθούμε και να τονίσουμε με το γεγονός ε, ότι χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη βιωσιμότητα. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα προωθήσει όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα όμως ο Χέλμουτ Σόλτς. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά τον εισηγητή γιατί μας εισήγαγε στην περιπλοκότητα του θέματος και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνειδητά ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, όπως είπαν ίσως και κάποιοι συνάδελφοι. Ε, μετεξελίσσοντας μια εμπορική στρατηγική. Τώρα είμαστε το 2018 του χρόνου, έχουμε ευρωεκλογέ. Και μένα με βασανίζει ήδη η ιδέα εάν η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στην εμπορική στρατηγική για όλους. Και αν μπορεί να διατηρήσει το όνομά του αυτό το πρόγραμμα, αν είναι ε, διαμόρφωση και τη θάσευση αυτή της παγκοσμιοποίησης. Λοιπόν, και κάποια άλλα στοιχεία, δύο τον αριθμό που με παιδεύουν πολύ. Πολύ συχνά ε, μπερδεύουμε, συγχαίουμε την παγκοσμιοποίηση με τη διεθνοποίηση παγκοσμιοποίηση είναι κάτι το αντικειμενικό που έχει να κάνει με την εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων και τη συνοδεύει και ταυτόχρονα εκφράζει ε, τις παγκόσμιες δομές παραγωγής αξίας. Και τίθεται το ερώτημα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση Κρατών είναι η ενδεδειγμένη δομή για να συμβαδίζει με αυτές τις εξελίξεις και να βάζει και ένα πλαίσιο. γιατί σε επίπεδο κατώτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνεται αυτό σε κρατικό επίπεδο. Έχουμε 12 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η ατζέντα και οι στόχοι ε, για την ανάπτυξη που είχαν συμφωνηθεί στη Νέα Υόρκη και μάλιστα να ολοκληρωθούν με επιτυχία. Απέχουμε πόρο από τη σοβαρή πρόθεση αυτών των θεμάτων. 17 είναι οι στόχοι. Πάνω από 140 τα προγράμματα, πολύ συγκεκριμένα. Αν τα δούμε αυτά, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα κράτη-μέλη, ε, οι κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια να ασχοληθούν με το θέμα. Τι θα κάνουμε για να είμαστε ρεαλιστικοί και σοβαροί στην αντιμετώπιση. Και στην έκθεση θα πρέπει να φέρεται περισσότερο αυτή η πολυπλοκότητα. Σήμερα απλώς το θίξαμε. Οπότε προβλέπω σε μια πολύ παραγωγική και συναρπαστική συνεργασία με τον εισηγητή και όλους τους κοιόδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως εταίρος ε, παραστά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, για να προχωρήσουμε σε άγνωστα εδάφη. Η κυρία Κιρτοντάλη. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά θα ήθελα να πω ότι όταν προτάθηκε αυτός ο διάλογος προέκυψε εξαιτία των δημόσιων διαδηλώσεων σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για το TTIP και τις διαπραγματεύσεις για την ΣΕΤΑ όταν χτυπάμε πόρτες σε πολλούς τομείς, όπως στη δικιά μου πικράτη, ε, ε, αυτός ο διάλογος γίνεται με ψηφοφόρους σε περιφέρειες οι οποίες έχουν θυχτεί από την παγκοσμιοποίηση και με θετικό και με αρνητικό τρόπο. πολλοί ήταν κοινικοί πάντα στην άποψη ότι οι παγκοσμίες ήταν πάντα κάτι θετικό, γιατί έβλεπαν τα αρνητικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες κοινότητες και τομείς και σε άτομα και ότι αυτά δεν λαμβάνονταν σοβαρή υπόψη από τους ε, πολιτικούς ηθήνοντες. Έχω προειδοποιήσει για όλα αυτά εδώ και πολύ καιρό και πολύ συναδελφοί μου και θεωρώ ότι η ψήφο για το Brexit και το ψηλό ποσοστό υπέρ του Brexit σε τη δική μου είχε να κάνει με την αντίδραση των ανθρώπων, των πολιτών ενάντια στις οικονομικές αλλαγές που συντελέθηκαν στις περιοχές παρόμοια δεν υπήρξε και σε περιοχές των ΗΠΑ, γιατί ο κόσμος ουσιαστικά δεν καταλάβαινε ότι ψήφιζε υπέρ ενό οράματο. Γι' αυτό αυτός ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός, γιατί έχει να κάνει με την πιστοσύνη στην εμπορική πολιτική, τις ε, δομές, ε, τις προστατικές δομές που θα πρέπει να υπάρξουν για αυτούς που έχουν εθιχτεί και όσον αφορά το greening και αυτά που ανέφερε ο σχεδόν συγκητής του EPP, στην αρχή της παρέμβασης συμφωνώ ότι οι εταιρείε θα πρέπει να είναι να... πρέπει να βάλουν λογοδοσία πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών και να υπάρχουν κανόνες για τις εταιρείε. Όμως δεν συμφώνησα με το συμπέρασμα ότι δεν έχουμε όλα τα πολιτικά εργαλεία που χρειαζόμαστε. Και υπάρχουν δύο παραδείγματα που είναι πολύ σημαντικά. Το ένα έχει να κάνει με το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε επιγόντω μία, ένα διάλογο για τη βιωσιμότητα, γιατί η αξιοπιστία των εμπορικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση τέθονται υπό αμφισβήτηση. υπό αμφισβήτηση. Υπάρχουν και παραβιάσει εργατικών δικαιωμάτων και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι υπάρχει ε, μια μεγάλη ευκαιρία σε εθνικό επίπεδο για ανάληψη ευθύνη. και είναι πολύ σημαντικό να να συμμετήσουμε ε, ένα μοσαϊκό από τις χώρες οι οποίες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε, όπω συμβαίνει στις, ε, στην Ολλανδία, στην Γερμανία για την υποχρεωτική εταιρική ευθύνη. Και θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε ίσες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε την παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να να αντιμετωπίσουμε τις ε, αλυσίδες εφοδιασμού σε επιχειρηματικό επίπεδο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την αναπαγκοσμιοποίηση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ. Για να συμφωνήσω με αυτά που προλαλήσατε, νομίζω ότι στους πολίτες δεν αρέσουν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Ε, μπορούμε να ακούσουμε πάρα πολλές καλές προθέσεις στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίηση, καθώς επίσης και τις αρνητικές συνέπειες μιας ε, ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης. Αυτή είναι μια θέση την οποία τηρούμε, την ακούσαμε, μετά από τις πολυέρθμες επικρίσεις που υπήρχαν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων, όπω η TTIP ή ε, αντίστοιχε. Υπάρχουν επίσης και κάποιες εμπορικές εμφανίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι υποδιαπραγμότευση. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει από τα λόγια στι πράξει. Το να λέμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και θα αντισταθμίσουμε την παγκοσμιοποίηση ενώ ταυτόχρονα διαπραγματευόμαστε κάποιες συμφωνίες οι οποίες ε, θα αρχίσουν να ισχύουν το 2019, το 2020 με αντίθετες συνέπειες από την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης, νομίζω ότι εδώ έρχονται τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που ακούνε οι πολίτες και οι πολίτες δεν μπορούν να ταυτιστούν πλέον. Δεν θέλουν να ανακόψουν την παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός οι πολίτες. Απλώς μας λένε ότι πρέπει να φροντίστε να προστατευτούμε. Και αυτό δεν σημαίνει προστατευτισμός. Προστασία σημαίνει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες για την παγκοσμιοποίηση. Όταν συναντούμε τις πολίτες, δεν είναι κατά του γεγονότο ότι προστατεύονται επενδύσεις. Αντιλαμβάνονται ότι όταν επενδύουμε ανά τον κόσμο υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία δεν ε, προστατεύουν επαρκώ τι επενδύσει. Το να υπάρχουν, για παράδειγμα, συστήματα όπω το ICS, το οποίο θέλει να προστατεύσει παγκοσμίω τι επενδύσει, λένε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όταν προσπαθεί κάποιο να φανταστεί ένα μηχανισμό προστασία των πολιτών για τα θεμελιώδη δικαιώματά του, της εργασίας ή των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, εδώ υπάρχει σπάνιδα απαντήσεων. Λέμε ότι θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να συζητήσουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις κλπ. Αλλά δεν θέλουμε να έχουμε μηχανισμούς κυρώσεων για την απώλεια αυτών των δικαιωμάτων. Θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε ε, δημιουργική για την προστασία των επενδύσεων. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τι προστατεύσουμε τι επενδύσει. Πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη δημιουργικότητα και για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των πολιτών και του περιβάλλοντο. Και εδώ και πάλι ακούμε δύο διαφορετικά πράγματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας λέει ότι τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξη έχουν κλείσει, αυτή είναι η θέση μας και τα ακούσαμε και σήμερα ότι δεν θα υπάρχει μηχανισμός κυρώσεων γιατί δεν είμαστε υπέρ ενός μηχανισμού κυρώσεων. Και αυτή η διπλή γλώσσα είναι αυτή η οποία δεν μπορούμε να αποδεχτούν οι πολίτε. Ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν στα πλαίσια τη συζήτηση να πάμε περαιτέρω, να μην έχουμε απλώ δηλώσει προθέσεων, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ήδη από σήμερα τις εμπορικές συμφωνίες ε, στις οποίες κάνουμε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών. Την κυρία Φενέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε που μας δώσετε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη σημερινή συνεδρίαση για ένα τόσο λεπτό ζήτημα για τις περιφέρειες και τις πόλεις μας. Ο κόσμος καταγράφει μια λιλεξάρτηση ανευπρεγουμένου. Αυτά ε, δεν μπορούμε να τα άρουμε καθημερινά και δεν θα ήταν και σωστή λύση. Κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργήσει περισσότερες ε, ζημιές ε, παρά ωφέλη. Επομένως πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η παγκοσμιοποίηση θα γίνει με έναν τρόπο με τον οποίο εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού επιθυμούμε. Και γι' αυτό η Επιτροπή των Περιφερειών ήδη έχει γνωμοδοτήσει δύο φορές για το έγγραφο προβληματισμό για τη διαχείριση της παγκοσμιοποίησης και για το εμπόριο στη συνέχεια και σήμερα έχουμε τη χαρά να συμβάλλουμε και ε, στις δικές σας τις απόψεις και άκουσα να υπάρχει ισορροπία από πλευράς από τον εισηγητή. Συμφωνώ απολύτως με την αρχική του παρέμβαση. Το νήμα λοιπόν που ενώνει ε, το σκεπτικό μας είναι να ε, διαφυλάξουμε την εδαφική μας κυριαρχία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την παγκοσμιοποίηση. Έτσι, στις συζητήσεις καταφέραμε να έχουμε μια πτυχή την οποία θα ήθελα να επισημάνω εδώ παρατηρητές στην ομάδα των εμπορικών συμφωνιών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να υποστηρίξετε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι και η άποψη των περιφερειών ε, μεταξύ των ε, σημείων διαπραγμάτευσης. Και επομένως να υπάρχουν και αξιολογήσεις εδαφικού αντικτύπου για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα ισχυρό μέσο και να βρούμε πριν από την έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας μιας εμπορικής συμφωνίας ποια είναι τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι συνέπειες για τις περιφέρειες και τις διάφορες περιοχές είναι πολύ διαφορετικές. Ορισμένες φορές είναι ε, καθοριστική σημασία για θετικά και άλλες φορές για αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε καλύτερες αποφάσεις, οι οποίες θα είναι θεμελιωμένες ε, ε, στο περιεχόμενο της συμφωνίας, να δούμε για παράδειγμα και τι γίνεται με τη στήριξη και να μην υπάρχει, ε, και, ή, άλλο να προλάβουμε τις ανετικές συνέπειες το να υποτιμήσουμε ή να ξεχάσουμε ότι κάποιες τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές οι οποίες προέρχονται από την παγκοσμιοποίηση, όπως πολύ σαφώς φάνηκε σήμερα από τη συζήτηση. Εμείς υποστηρίζουμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να αποτρέπουν στις ε, ε, δημόσιες διοικήσεις οποιοδήποτε επίπεδο να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες και να διευρύνουν και το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν και να προβλέπουμε και συγκεκριμένες κοινωνικές ηλικίε Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα. Όπω επίση είναι σημαντικό να προβλέψουμε και την ικανότητα επενδύσεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ώστε να είναι και πιο ευέλικτη η διαδικασία αντιμετώπιση τη παγκοσμιοποίηση. Και τέλο, δύο πολύ σημαντικά για μας σημεία, τα οποία αφορούν και τη συζήτηση σε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητούμε τώρα και αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι η εδαφική συνοχή και η χρηματοδότηση χωρίς αλλαγές των μέσων για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικά και φυσικά θα πρέπει να προσαρμοστούν και στο περιεχόμενο αλλά και τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν, κυρίως τα προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα. Μια δεύτερη πτυχή που είναι πολύ σημαντική για μας και για την οποία ανησυχούμε πολύ είναι το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο γι' αυτό, ενώ είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ στεναρή πρόταση από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για αυτήν ακριβώς τη πτυχή σα ζητούμε να σταθείτε στο πλευρό μας. Γιατί θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος για να απαντήσουμε, αν και με πιο ευέλικτο και προληπτικό τρόπο, σε κάποιες από τις κοινωνικές ανισότητες, ε, τις οποίες έθιξαν και οι συνάδελφοι προηγουμένω. Για παράδειγμα, η Αγγλίδα συνάδελφος που αναφέρθηκε στο Brexit. Και αυτό ε, τονίστηκε δεόντως εδώ. Έχουμε συλλογική ευθύνη να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτούς που θα μπορούσαν ε, να πληγούν αρνητικά ή που έχουν ήδη πληγεί με αρνητικό τρόπο. Και θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο εάν κλείσουμε τα μάτια σε αυτές τις περιοχές, τομείς και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό. Για όλα αυτά σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε βεβαίως εξαιρετική ε, δουλειά. Ευχαριστώ ε, για την the τη Επιτροπή ο Λούκα Κάρλι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή και τα αξιότιμα μέλη που εξέτασαν τι απόψει του. Όπω θα θυμάστε, αυτό το έγγραφο για την αξιοποίηση τη παγκοσμιοποίηση εκδόθηκε ε, την περίοδο του State of the Union μαζί με άλλες προτάσεις. Δεν είναι στρατηγική ε, συνεχίζει τις βασικές αρχές του Trade for All, εμπόριο για όλους και ε, δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέσσερις βασικές ιδέες ε, τις οποίες θα αναφέρω εν συντομία. Η πρώτη είναι ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αντίθεση με τον κύριο Τραμπ ότι οικονομική το οικονομικό άνοιγμα είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των ε, πολιτών συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις ε, ε, σε τη το και με την Αυστραλία και με την Νέα Ζηλανδία. Υπήρξε και ένα βασικό μήνυμα από τον κύριο Γιούγκερ ότι δεν είμαστε αφελεί όσον αφορά το οικονομικό άνοιγμα. Θα πρέπει να υπάρχουν ίσε ευκαιρίε και ένα συγκεκριμένο ε, πλαίσιο αμοιβαιότητα. Υπογνωσμή για την ανάγκη να ολοκληρώσουμε τη νέα μεθοδολογία για την Κίνα, για το anti-dumping την παρακολούθηση των ξένων επενδύσεων, να ολοκληρώσουμε τις νομοθετικέ προτάσεις όσον αφορά ε, το μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις. Το δεύτερο είναι το Trade for All, είναι οι αξίες οι οποίες είναι ο ακρογωνίος λήθο για την πολιτική μας, δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική, αλλά χρησιμοποιούμε την οικονομική πολιτική για να προωθήσουμε τι αξίε μα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αξιοποίηση τη παγκοσμιοποίηση μα δίνουν την εντολή να διαπραγματευτούμε σε πολυμερέ επίπεδο. Είχαμε μια μακροσκελή συζήτηση για το πώς θα αλλάξουμε την παιδική μας πολιτική με το πολυμερές δικαστήριο επενδύσεων. Έτσι διεξάγουμε την οικονομική πολιτική και κάναμε ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τη διαφάνεια. Θυμάμαι με Έλληνε να αναφέρουν ότι η εμπορική πολιτική συμβαίνει και των θυρών. Ταυτόχρονα σε αυτήν την ανακοίνωση ανακοινώνουμε την πρώτη τη Επιτροπή για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Είναι ένα βήμα άνευ προηγουμένου το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερη διαφάνεια κάτι που δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη ε, περίπτωση σε σχέση με διεθνεί σχέσει. Επίση, η ενίσχυση των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων για να συμμετήσουν τη δικιά του ε, γνώμη και να ακουστεί η φωνή του μέσω τη κυβέρνησή του ω προ το πώ θα του επηρεάσει αυτή τη συμφωνία στο μέλλον. Και αναφέρω τα Εθνικά κοινοβούλια, γιατί προκύπτει και ένα τρίτο μήνυμα από αυτή την ανακοίνωση, γιατί αν η Ευρώπη θέλει να προσπαθήσει να εξοπλίσει την παγκοσμιοποίηση, και να γνωρίσει το μέγεθος αυτής της απόπειρα, θα πρέπει να ρωτήσουμε ε, και η γνωμοδότηση της Συγκαπούρης μας δίνει μια γερή βάση. Φυσικά η πολιτική διαδικασία θα συμπεριλάβει και τις τοπικές κοινότητες, περιοχές και το εθνικό επίπεδο, αλλά η διαδικασία της λήψης αποφάσεων για τα καθαρά θέματα εμπορικής πολιτικής χρειάζεται νομιμότητα και αυτή αυτό επικαιρώνεται μόνο μέσα, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέσω των εθνικών κυβερνήσεων που θα ε, παρουσιάσουν τις δικές τους ε, τοποθετήσεις. Τέλος, είναι εύκολο να μιλάμε αλλά πρέπει παράλληλα να δείχνουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε και αυτά που προσχόμαστε. Αυτή λοιπόν η έκθεση ε, συνοδεύεται από μια έκθεση εφαρμογής στην οποία δείχνουμε τι έχουμε πράξει μέχρι στιγμής και τι παραμένει να γίνει. Δύο τελευταία σημεία, κάποιος ανέφερε για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, είναι προ, ε, ε ένα κομμάτι του MFF. Προτείνεται μία αύξηση, έχει να κάνει με τα διευθυντικά ταμεία που παρέχουν ε, ανθεκτικότητα, η οποία δεν προέρχεται μόνο από ε, το εμπόριο, αλλά και από ε, την αλλαγή στη τεχνολογία, στην κοινωνία, από εξωτερικέ και εσωτερικέ πιέσει. Το γνωρίζουμε όμω καλά το θέμα και δίνουμε προτεραιότητα σε αυτό. Επίση, για τον πόρο και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι και αυτό ένα σημείο σημαντικό. Πιστεύουμε από την πλευρά μα και το έχουμε στις πολλέ φορέ αυτό το θέμα ότι ε, πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις και θεωρούμε ότι μέσω της προσέγγισής μας και του διαλόγου και της δημόσιας πίεσης που θα ασκηθεί συν τα 15 σημεία για την άσκηση πίεσης ε, στην ενδιαφέρον Αμερική και στους εταίρους θα πετύχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λοιπόν σαφές σε αυτό το τελευταίο σημείο ότι έχουμε μεγάλες διαφορές. Και κατά δεύτερον διαδικασία δεν ήταν κατάλληλη για να σεβαστεί το Κοινοβούλιο, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Παρουσιάστηκε ένα έγγραφο, ακόμα και στο Συμβούλιο, μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση. Δεν είναι κατάλληλος τρόπος αυτός και όσον αφορά το περιεχόμενο, τα 15 σημεία μπορείτε να τα εφαρμόσετε άμεσα. Μπορείτε να το έχετε κάνει πριν από πέντε χρόνια αυτό. Άρα δεν υπάρχει πραγματική πρόεδρο, πρόοδος είναι μια απόφαση της Επιτροπής ενάντια πολλών που παρευρίσκονται εδώ. Και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα για μια μελλοντική μη συνεργασία. Και το έχουμε λάβει το μήνυμα αυτό. Πολλοί συνάδελφοι εδώ. Ιωάχιμ, ο λόγος εσένα. Ίσως θα έπρεπε να πω ξεκάθαρο σαν αφορά την Επιτροπή και αυτά πάνε στο 2017, σήμερα έχουμε περισσότερε πληροφορίε. Και θεωρώ ότι οι συνεισφορέ των σκιωδών να δημιουργήσουν μια πολύ καλή βάση για διάλογο, γιατί υπάρχει συμφωνία ότι ως προς τις ε, ως προτερήματα της ε, παγκοσμιοποίησης του υπήρξε εξέλιξη στο παρελθόν και ότι υπάρχει ενότητα αλλά και υπάρχουν και προκλήσεις και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη έχει να κάνει με τους ε, στόχους, ε, τη βιωσιμότητα της και οι στόχοι τη συμφωνία των Παρισίων. Το δεύτερο θέμα που θέλω να συνδέσω και θεωρώ ότι θα υπάρξει ένας ε, διάλογος πάνω σε αυτό, αφορά την πολυπλοκότητα θα μας που ο συνάδελφο Σόλτ. θα πρέπει να υπάρξουν διεθνεί κανόνε, Αυτή είναι μια πρόκληση πρόκληση. Από την πλευρά είναι αυτά που θα θέλαμε εμεί να γράψουμε και αυτά που μπορούμε να γράψουμε, γιατί υπάρχουν και άλλοι παίκτε σε παγκόσμιο επίπεδο που ενδεχομένω βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Ο Τραμπ φυσικά και δεν συμφωνεί μαζί μα. Όσον αφορά τον προστατευτισμό ε, του Τραμπ, αυτό είναι κάτι που το αρνούμαστε. Είμαστε υπέρ τη ανοιχτή οικονομία, αλλά πώ μπορούμε αυτό να το διαμορφώσουμε τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, πώς θα ενισχυθούμε, ποιες είναι οι αποστολές μας ως προς ε, την ε, βιωσιμότητα. Δεν έχουμε ε, πρώτη προτεραιότητα την βιωσιμότητα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πώς το δικό μας το εμπόριο μπορούμε να το συνδέσουμε με την βιωσιμότητα. Τι κάνουμε στην εμπορική πολιτική, όταν σε πολλές περιπτώσεις δυσχεραίνουμε τη βιωσιμότητα. Θα πρέπει να δώσουμε στρατηγικές απαντήσεις, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έκθεση, για να ξεκινήσουμε το διάλογο. προ τι ανησυχιώδεις συζήτητες, πολλούς, ε, πολλά άλλα σημεία και άλλε προσεγγίσεις και θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο βήμα θα είναι ο διάλογο για το σχέδιο γνωμοδότησης Σημείο 10. Γενικός προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τμήμα που αφορά το εμπόριο. Χαίρομαι που βλέπω τον εισηγητή της Επιτροπής Προπολογισμών. Ε, Βιώτη. Τον κύριο Βιώτη. Θα του δώσω μέσω στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία εδώ σήμερα στην Επιτροπή σας σχεδόν στο τέλος ε, μιας μακριάς περιοδίας που έκανα σε όλες τις εξειδικευμένες επιτροπών που, επιτροπές που κάνω αυτές τις εβδομάδες και ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές για μένα αυτές οι επισκέψεις ε, και αυτές οι συναντήσεις ε, διότι από πλευράς της δικής σας καταλαβαίνω κάποια πράγματα τα οποία είναι απλώς αριθμοί στον προϋπολογισμό αλλά πολύ συχνά δυσκολεύομαι να καταλάβω την πραγματική του σημασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ λοιπόν αυτέ οι συναντήσεις για μένα. Πολύ σύντομα, διότι η σημασία αυτή τη συνάντηση είναι περισσότερο να ακούσω την Επιτροπή σα και τα προβλήματά σα. Ε, δύο στοιχεία τα οποία θα ήθελα να σα πω όμως ε, καταρχήν. Ε, όσον αφορά τη μέθοδο, η πρόθεσή μου είναι όπως έκαναν και οι συνάδελφοι τα προηγούμενα χρόνια, να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση ε, για τη δουλειά που πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον προπολογισμό, όχι μόνο από πολιτική σκοπιά, ε, επομένω ε, όχι μόνο λαμβάνοντα υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερε πολιτικέ ομάδε, αλλά και από θεσμικό πλέ, ε, επίπεδο. Δηλαδή να έχουμε στήριξη από όλε τι επιτροπέ και στη στάδια του, στα στάδια του τριμερούς και, διαλόγου συγγνώμη, και στην συνδιαλλαγή και θα ήθελα να ακούσω και τι προτάσεις ε, έχετε να μου κάνετε, ε, γνωρίζοντας ότι αύριο υπάρχει και μια πολύ σημαντική ψηφοφορία για την μακροοικονομική βοήθεια για την Ουκρανία και μάλιστα με ένα πολύ σημαντικό ποσό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εμείς σήμερα μιλούμε χωρίς να έχουμε ακόμα τον προϋπολογισμό και το προσχέδιο προπολογισμού από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 23 Μαΐου. Υποχρεωτικά λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να δούμε ακριβώς κάθε αριθμητικό στοιχείο, αν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις είτε θετικές είτε αρνητικές. Τώρα είμαι εδώ για να τίνω ευήκο νους στις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο, ο κύριος Δάρτμουθ. Μεγάλο προνόμιο να ε, παίρνω το λόγο. Σπάνια ακούτε πολιτικούς να σας λένε ότι ήρθα για να σας ακούσω. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να πω ότι το ε, εκτιμούμε σφόδρα αυτό. Δεν ε, Βλέπω πολλούς βουλευτές εδώ. Κοιτάξτε, έχω γράψει ένα βιβλίο το εμπόριο, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πολύ, εκτός από την εκπρόσωπο του ΙΣΙΑ. Ε, δεν γνώρισε μεγάλη ε, απήχηση. Θα ήθελα να έχει κυκλοφορήσει <laughs> περισσότερα αντίτυπα. Για το εμπόριο, λοιπόν, ε, για τη γνωμοδότηση. Θα πρέπει να τονίσουμε την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα γνωρίζουμε πλέον στη δεκαετία του 70 δεν ήταν σαφές αυτό, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ηγούνται στην οικονομία, την καθοδηγούν, δεν την ακολουθούν. Εκείνες ε, παράγουν ε, ανάπτυξη, μεγένθηση και καινοτομία και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η μακροοικονομική βοήθεια είναι κάτι που θέλει διευκρίνηση. Τι συμπεριλαμβάνει εκεί ο προϋπολογισμός. Συμπεριλαμβάνεται και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο που θα αποχωρήσει. Ξέρετε ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό για την βοήθεια, για την αναπτυξιακή βοήθεια. Α, πόσο χρόνο έχω. Ε, α, δεν πειράζει, γιατί συνηθίζω να τηρώ το χρόνο. Είναι πραγματικά τεράστιος ο προϋπολογισμός μας για την ε, οικονομική βοήθεια. Ε, και ποιο είναι το κλάσμα που πηγαίνει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και πώς έχετε κάνει τους υπολογισμούς σας για την περίοδο μετά το Μάρτιο του 2019. Η γνωμοδότηση που προτείνω εγώ τι λέει ότι η μακροοικονομική βοήθεια θα πρέπει να προσανατολίζεται με βάση τις ανάγκες και όχι τις πολιτικές. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και μια ενίσχυση που συνδέεται με το εμπόριο. Aid for trade λέγεται αυτό. Δίνουμε βοήθεια για να κάνουμε εμπόριο. Εγώ θα προτιμούσα trade, not aid. Εμπόριο, όχι βοήθεια. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτό να ασχοληθεί. Τώρα, σε εμπορικέ συμφωνίες Ποιο είναι το ενδιαφέρον. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα στατιστική, αν δείτε όλες τις εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να διαβάσετε κάτι ενδιαφέρον. Το ΑΕΠ των χωρών αυτών με τις οποίες έχουμε εμπορικές συμφωνίες, αν το διαβάσετε, μόνο εννέα από αυτές έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ από τη Δανία και καμία μεγαλύτερο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ιαπωνία, ας πούμε, θα δει την ε, συμφωνία της να ε, ολοκληρώνεται προσεχώς και θα αλλάξει αυτό κατά ε, μία ποσοστία μονάδα. Τι προτείνω λοιπόν εγώ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, όσο και αν είναι επιθυμητά, ε, δεν είναι ο χώρος τους οι εμπορικές συμφωνίες. Τουλάχιστον αυτή είναι η εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, απορρίπτω την άποψη που λέγει ότι το εμπόριο θα πρέπει να είναι ένα... Μάλλον, ε, πρέπει να είναι εργαλείο ε, δημιουργίας, ανάπτυξης, ευημερίας και θέσεων απασχόλησης και όχι εργαλείο εξωτερικής πολιτικής για αλότριους σκοπούς μόνο για το ε, εμπόριο θέλω να μιλήσω και τώρα μας βίνουν τα φωτά και τελειώνει ο χρόνος μου. Ο ευρωπαϊκός προπολογισμό θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι αλλάζουν τα ε, οικονομικά δεδομένα με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και θα πρέπει να αυξηθεί η συνεισφορά των άλλων κρατών μελών που θα δυσκολεύσει σοβαρά διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, κάποια κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεσμεύονται από τη συνθήκη να έχουν περιορισμένα ελλείμματα στον προπολογισμό τους. Άρα, όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει τον προπολογισμό της και όχι να τον αυξήσει. Και μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι η μεγαλύτερη οικονομία που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχει μία έδρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι δύο. Και υπάρχει και μια τεράστια ανομαλία θα συμφωνήσουμε όλοι, με εξαίρεση ένα μέλλον της επιτροπή Το Λουξεμβούργο είναι μακράν η πλουσιότερη χώρα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με, ε, μεταξύ των έξι πλουσιότερων ε, χωρών στον κόσμο. Έχουμε όμως 2.000 υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο. Μήπως να τους πάμε στη Νότια Ιταλία ή στη Βουλγαρία που είναι φτωχή χώρα να μετεγκατασταθούν εκεί να μετεγκατασταθούν. Δεν έχει καμία έννοια να είναι στο Λουξεμβούργο. Καλά. Αμφιβάλλω αν όλα αυτά που σας λέω θα βγουν ως γνωμοδότηση από την Επιτροπή ΙΝΤΑ, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό και στην ευκαιρία να τα πω. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που με ακούνε τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Έξι λεπτά της δόξης σας. <laughs> Uh, λοιπόν, οι σκιώδες τώρα. Ο κύριος Φιάλνερ απουσιάζει, η κυρία Ανδρική Ένε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος του Κρίστοφ Φιέλνερ, συναδέλφου από το ΕΛΚ και σκιώδους εισηγητού Γι' αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που συζητούμε σήμερα. Πάρα πολύ λίγα σχόλια. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει την υποκείμενη ε, αρχή ε, και τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2019. Σίγουρα θα πρέπει κατά προτεραιότητα στόχος ε, να είναι η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου ε, των πολιτών μας για να υποφεληθούν από την παγκοσμιοποίηση. Αυτό σημαίνει επένδυση στην έρευνα ε, και την καινοτομία έτσι ώστε οι οικονομίες μας να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική, θα πρέπει να έχει τους απαραίτητους πόρους στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δίνει συνέχεια στη φιλόδοξη ε, στρατηγική της και να μπορούν οι εταιρείε να κάνουν πιο εύκολα εμπόριο, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, για να, για να συμμορφώνονται καλύτερα με τους κανόνες ε, προέλευσης. Αυτά σε γενικές γραμμές και προσβλέπουμε να δούμε και το σχέδιο της νομοδότησης για να έχουμε και μελλοντικές συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστέ και δημοκράτε, η κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ντανιέλε, που ακούς όλες τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας και ελπίζουμε ότι οι υποδείξεις μας τουλάχιστον θα συμπεριληφθούν ε, στη συλλογική έκθεση και πραγματικά η σκέψη μας ε, είναι λίγο διαφορετική από αυτήν ε, που παρουσίασε ο εισηγητής κάποιες σκέψεις. Εμείς θα παρουσιάσουμε ως ομάδα τις προτεραιότητές μας, οι οποίες ε, δεν διαφέρουν και πολύ από αυτές που είχαμε παρουσιάσει πέρσι, διότι θεωρούμε ότι αν η παγκοσμιοποίηση ε, πραγματικά δεν πρέπει να αφήσει κανέναν πίσω, όπως αυτό ε, είναι αυτό που πιστεύουμε, πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη διάταξη μεταξύ των πολιτικών και πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να υπάρχουν και στοιχεία από άλλες επιτροπές ε, που έχουν σχέση και με την επιτροπή μας ε, και με την οποία είμαστε σε συνεχή επαφή. Δεν θεωρούμε ότι μία εμπορική συμφωνία από μόνη της μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Πρέπει λοιπόν να ε, προσθέσουμε και μία σειρά μέσων χρηματοδότησης που έχουν αυτό το σκοπό. Τα τρία σημεία λοιπόν, τα τρία βασικά σημεία για μας είναι καταρχάς να ξανασκεφτούμε εις βάθος το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση διότι κατά την άποψή μας δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό, να μπορεί να παρέμβει όχι μόνο ε, σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει μια κατεπίγουσα ανάγκη, μια κρίση, αλλά να είναι και σε θέση να βρει μέσω συντονισμού με αναλύσεις επιπτώσεων που ε, μπορούμε ενδεχομένως ε, να έχουμε ανάπτυξη να έχουμε όχι τόσο μια προληπτική δράση, αλλά να μπορεί να παρέμβει ε, στα σπάργανα μιας κρίσης. Ε, δεύτερον, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυξήσουμε τα κονδύλια τα οποία αφορούν ε, την ε, ε διαπραγματευμένωση εμπορικών συμφωνών, γιατί είδαμε και με τις χώρες ΣΑΚΕ ή με την Κορέα, Κορέα ότι είναι ψευδέστηση να ζητάμε, για παράδειγμα, να συμπεριληφθούν και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, αν δεν υπάρχει αποτελεσματική του χρηματοδότηση. Και διαπιστώσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για όλες τις πτυχές που αφορούν την παρακολούθηση, αλλά και να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η εμπορική συμφωνία στο σύνολό της ε, και στις οικονομικές πτυχές. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμείνουμε ε, όσον αφορά τις αυξήσεις αυτές. Ε, τέλος, ε, πέρσι, εγώ με την συνάδελφο Εμακολάδα Ροντρίγκε παρουσιάσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για συλλογή στοιχείων που αφορούν ε, την ισότητα των φύλων και φέτος θα θέλαμε να προτείνουμε κάτι στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας που ελπίζουμε να τύχει και ευρεία υποστήριξη και να έχει στόχο την ενδυνάμιση του προγράμματος Regiotex. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Μακλάρκεν. Ο κύριος Λούνες κανονικά θα μιλούσε για αυτό το θέμα, ε, για τον προπολογισμό, θα πλαίσια της Ίνταλα. Η ομάδα μας δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να ε, εγγράψουμε κονδύλια στον προπολογισμό, να προβούμε σε ανάληψη υποχρεώσεων δηλαδή κλπ. Ε, πριν λυθεί το θέμα με το backlog, της, της πληρωμέ πληρωμές και της ε, κληρονομίας του παρελθόντος. Συμφωνώ με το συντάξει νομοδότηση για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την καινοτομία και πραγματικά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις προτεραιότητες στα κονδύλια του προπολογισμού. Αντί να ζητάμε συνέχεια όλο και πιο πολλά λεφτά. Άλλος. Α, ο κύριος Κέλλη. Ε, πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Τα σχόλια του συναδέλφου και καλού φίλου Ντάρθμου θα βρήκα ε, ενδιαφέροντα κατά τα άλλα, αλλά θέλω να πω το εξή. Αυτό που είπε και ο συνάδελφος Βιώτη για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Πραγματικά πρέπει να είναι μεγαλύτερο το ταμείο αυτό και να καλύπτει περισσότερες παραμέτρους από ό,τι ισχύει σήμερα για να αντιμετωπίζουμε κάθε είδους ε, κρίση που μπορεί να βρούμε μπροστά μας. Και αυτός είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπόνια μας στους πολίτες όταν υφίστανται τα πάνδυνα και έχουν τέτοια πικρή ανάγκη. Μέχρι τώρα δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό λόγω των περιορισμών και των κανόνων, αλλά και του προπολογισμού του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση. Και αν συζητάμε για αυτό το θέμα, που το κάνουμε ιδιαίτερα στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επόμενο προπολογισμό, για το διπλασιασμό των κονδυλίων για το Εράσμου και διάφορα άλλα τέτοια ε, πολύ αξιέπαινα. Αλλά θα πρέπει να δούμε Πού είναι ο κόσμος που ειναι ο κόσμο που περναει τη μεγαλύτερη δυστυχία και συμφορά είναι όταν χάνει τη δουλειά του ή όταν έρχονται διάφορε θεομηνίε στο κεφάλι του και θα πρέπει ε, γρήγορα και με τον κατάλληλο τρόπο να απαντούμε. Και αυτό γίνεται μόνο όταν έχει ένα προπολογισμό που σου επιτρέπει να το κάνει. Πολύ σημαντικό. Το είπε μια συνάδελφο, η κυρία Μόσκα προηγουμένω και συμφωνώ μαζί τη. Ευχαριστώ. Η Χάιντι, Χάουταλα. Ε, ε, αυτό να κηρύσουμε σκιώδη συγκήτρια. Ε, δύο πράγματα πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αξιοποιήσουμε τα προγράμματα Aid for Trade, ε, βοήθεια για το εμπόριο. Έχω μια μεγάλη παράκληση να υποστηρίξουμε τις γυναίκες που ε, είναι παραγωγοί, που ιδρύουν επιχειρήσεις και μπαίνουν και στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής ε, πλούτου. Αφού γίνεται πια τόσος λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τους απαραίτητους πόρους ε, και υπαλλήλους για να οργανώνει όλα τα προγράμματα και τα πιλωτικά προγράμματα να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι. Εκεί χρειάζεται λίγη βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία αυτά ε, το Aid for Trade, βοήθεια για εμπόριο, για να δημιουργούνται ικανότητες στις άλλες χώρες, υποσαχάριες και τα λοιπά. Πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά είναι και ένα μέσο αυτό υποστήριξης ε, συστημάτων δικαίου εμπορίου. Και πραγματικά θέλουμε πολύ να ενισχυθεί. Ακούω διάφορες φήμες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει περικοπές στο Aid for Trade υπέρ του νέου αυτού συμφώνου για τη μετανάστευση. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Ισχύουν αυτά. Αληθεύουν. Γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στο πρόγραμμα Aid for Trade. Είναι και μήνυμα προς τον κύριο Βιώτη. Είναι σημαντικό το μέσο αυτό για δίκαιο εμπόριο μην το πειράξουμε. Ο Πίτερ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τον συντάκτη γνωμοδότησης της Επιτροπής σας που αναφερθήκατε στα θέματα του προλογισμού. Είναι πολύ επίκαιρο να συνδέεται τη συζήτηση ε, για την παγκοσμιοποίηση με τον προπολογισμό είναι ωραίος ο τρόπος που έχετε έτσι, καταρτήσει την σημερινή ημερήσια διάταξη, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και έχει σχέση ο προπολογισμό και με τη διθάσευση της παγκοσμιοποίησης. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι ένα σημαντικό μέσο και εργαλείο για να ε, βοηθήσουμε να έρθει ανάπτυξη, θέση εργασίας, να βοηθήσουμε ε, την ανάπτυξη και είναι σχετικά φθηνό μέσο για να το κάνουμε αυτό σε σχέση με όλο τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εμπόριο δεν ε, επιβαρύνει ιδιαίτερα τον προπολογισμό. Για τα ε, συγκεκριμένα θέματα που αναφέρετε, μερικές μόνο αντιδράσεις. Πρώτον, βοήθεια για το εμπόριο H4 Εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιε φήμε, Πρόεδρε, όπω αυτέ που ακούτε εσεί, για ενδεχόμενε αλλαγέ στον προπολογισμό. Και είναι δύσκολο να αποφανθεί κανεί ε, πριν αποφασίσει για τα ποσά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άλλη εβδομάδα. Σε σχέση με τα όσα είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ρόλο τους, ορισμένοι από σας, και τα ε, μέσα που έχουμε, εμείς μπορεί να έχουμε ένα μετροπαθή ε, προϋπολογισμό, αλλά προς τα εκεί στρεφόμαστε και θα διερευνήσουμε και τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν, να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταλάβουν καλύτερα τους κανόνες προέλευσης. Επίσης, με άλλα πιλωτικά προγράμματα και με την Επιτροπή σας, ε, είχαμε τη δυνατότητα να ενημερώνουμε καλύτερα τον κόσμο και να φτάνουμε σε αυτό. Mentioned, uh, very... Όπως είπατε επίση, είναι σημαντικό να έχουμε κοινή απάντηση από διάφορες πολιτικές ε, στην αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης και από τα διαρθωτικά ταμεία δηλαδή και από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ε, που είπε ο κύριος Κέλλη και ε, σε προηγούμενη συζήτηση θυμήσαμε ότι προτείνει αύξηση κατά 15% ε, στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. Ε, ε, κυρία Μόσκα και άλλοι, μιλήσατε για την υποστήριξη της συμμετοχής κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα στις δομές που δημιουργούμε στις εμπορικές μας συμφωνίες για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμβουλευτικά όργανα, αλλά και χρηματοδότηση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Πάντα το κάνουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό για να εξηγούμε την εμπορική πολιτική και να την ε, προάγουμε. Τα υπόλοιπα σχόλια τα σημειώνω και περιμένουμε ενδιαφέρον τη συνέχεια που θα δώσετε στη συζήτηση αυτή. Και χαίρομαι για τα καλά σας λόγια και την υποστήριξη για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Πάντα θα πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να κάνουμε τη δουλειά που εσείς χρειάζεστε και, και η Ευρώπη φυσικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σχόλιο από την Επιτροπή Προπολογισμού. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Όπως ε, πολύ σωστά φανταζόμουν, είναι πάντα χρήσιμο να συμμετέχει κανείς ε, στις εξειδικευμένες επιτροπές, διότι μου διευκρινίσετε κάποια στοιχεία, όπως είπα και στην αρχή, και θα ήθελα τώρα να σταθώ σε τρία στοιχεία. Πρώτον, οι εκκλήσεις που έγιναν ε, σε όλες τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να σας πω ότι αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο λαμβάνω από όλε τις επιτροπές και είναι κάτι επί του οποίου μπορώ να πω ότι ε, υπάρχει ε, σύμπτωση απόψεων από όλα το κοινοβούλιο. Ο καθένας βέβαια στον τομέα του, ε, καστο στο είδος του, αλλά ε, πρέπει να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και αυτό είναι βαθιά ριζωμένο σε όλο το κοινοβούλιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κάτι το οποίο επαναλάβατε αρκετέ φορές. Εγώ ασχολούμαι συχνά με αυτό στην Επιτροπή Προπολογισμών, διότι ούτω ή άλλω από εκεί περνάει εν τέλει, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στον προπολογισμό του 2019. Ε, το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι άλλη συζήτηση. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει και γι' αυτό, όπως και για άλλα, μια γενική μεταρρύθμιση και ελπίζω όπως και εσείς ότι, όπως είπε και η Αλέσια αλλά και ο συνάδελφος Κέλλη, να πάει προς την κατεύθυνση της ε, διεύρυνσης του προπολογισμού και να μην ε, έρχεται κατόπιν εορτής ε, στις κρίσεις που συνέβησαν, όχι να τις προλαμβάνει, αλλά να είναι στο πλευρό των κρατών μελών και να έχει σημαντική πρικοδότηση. Αυτό βέβαια θα το δούμε με το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα το δούμε και στο τέλος του, του, του σχεδίου προπολογισμού. Τώρα θα δούμε και τι γίνεται με το ε, συνέπειες του Brexit στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Να δώσω ίσως άσχημη είδηση στον συνάδελφο Ντάρκμουθ, αλλά πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκε και για το 2019 και το 2020 να συμβάλλει στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, για τον προπολογισμό για τον οποίο είμαι αρμόδιος εγώ, μπορούμε να είμαστε ήσυχοι για το έτοιμά σα τώρα για το μέλλον να μειωθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωση, Είδαμε στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρά το γεγονός ε, ότι δυστυχώ λέω εγώ, θα γίνουμε 28-27, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση, αν και μικρή λοιπόν, εγώ ελπίζω να είναι και μεγαλύτερη, θα υπάρχει αύξηση του ε, προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, και πριν ε, κλείσω κάτι τελευταίο. Όπως είπα στην αρχή, σε όλες τις άλλες επιτροπές, ε, πρόθεσή μου είναι να προχωρήσω σταδιακά. Να μην λύσουμε τώρα με μια συνάντηση ε, και τα θέματα σχέσεις μεταξύ Επιτροπής ΣΥΝΤΑ και Επιτροπής Προπολογισμών, αλλά είτε άτυπα είτε επισήμως ε, να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα τα επόμενα στάδια της εξέλιξης του προπολογισμού από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντάρτμαου. Θέλετε να προσθέσετε. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για όλα αυτά που είπαν και το οποίο θα τα λάβω υπόψη. Και επιπλέον να ευχαριστώ τον καλεσμένο μας. Ήταν πολύ, ήσασταν πολύ σύντομος. Ευχαριστώ. Καλή τύχη με τον προπολογισμό. Έτσι φτάνουμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Επενδύσεων. Αρχικά θεώρησε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια ανακοίνωση γι' αυτό. γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις. Το τελευταίο μήνα. Λοιπόν, έχουμε την πρόταση ενός πολυμερούς δικαστηρίου επενδύσεων, κάτι που υποστηρίχθηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υιοθέτησε μια οδηγία διαπραγματεύσεων. Άρα τα πράγματα έχουν τεθεί σε κίνηση. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί και φυσικά να δούμε τι σημαίνει αυτό στις, για τις διμερείς συμφωνίες εμπορίου. Το δικαστικό σύστημα με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, και το Μεξικό σχετικά με τι επενδύσεις ποια, είναι ο συσχετισμό, ποιε είναι οι σχέσει. και μετά διάβασα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για κάποιες διμερείς συμφωνίες με το ISDS σύστημα που είναι παλιό και η απόφαση ήταν ότι δεν είναι σύμφωνος αυτές τις συμφωνίες με, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα. από όσο καταλαβαίνω σε αυτή τη μεταρρυθμιστική διαδικασία δεν θα είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε άλλη μια φορά για ένα μηχανισμό ASDS. Και ενδεχομένως το πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα όπως άκουσα από τη βοηθό μου πριν από λίγες μέρες είναι ότι μετά την ε, υιοθέτηση του κανονισμού του 2012 η Επιτροπή συμφώνησε να υπάρξουν διμερείς συμφωνίες επενδύσεων και πολλά κράτη-μέλη το έπραξαν αυτό σύμφωνα με το πρότυπο SDS. Είχαμε δύσκολες συζητήσεις με αρμόδιους της Επιτροπής, ακόμα και με επίτροπο για το σύστημα επενδύσεων. Ήταν κάτι παράδειγμα αυτό που συνέβη για μένα. Έχουμε αυτή τη διμερή συμφωνία ε, επενδύσεων μεταξύ των μελών, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή. Πώς έγινε αυτό. Μια ερώτηση που θα ήθελα να απαντηθεί. Τέσσερις ερωτήσεις που θα ήθελα να απαντηθούν. Και κάποιες εξηγήσεις από τον Κάρλο Πετινά. Θα τις προτιμούσα γραπτές τις απαντήσεις. Παρακαλώ, μπορείτε να ξεκινήσετε. Thank you, Chairman. Um, very Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, όντως. Και με χαρά να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα λίγα λεπτά που έχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όπως σας έχουμε πει και το κατά το παρελθόν, από το 2015, από τότε που εγκρίναμε ένα σύστημα ε, συνολικής μεταρρύθμισης της επενδυτικής μας πολιτικής, έχουμε επιτύχει ένα σημαντικό αριθμό διαπραγματεύσεων. Σημαντικές διαπραγματεύσεις δηλαδή που καταφέραμε να εντάξουμε το νέο σύστημα τη νέα μέθοδο, τη μεταρρυθμισμένη. Τι σημαίνει αυτό, η αναθεωρημένη μέθοδος. Είναι πιο σαφής η διατύπωση των διατάξεων ε, για την προστασία των επενδύσεων και ε, χωρίς να επιδέχονται υπερβολικές ερμηνείες και το σύστημα των επενδυτικών ε, δικαστηρίων. Πρόσφατα παρουσιάσαμε τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με προστασία επενδύσεων. Βεβαίω η ΣΕΤΑ είναι μια συμφωνία με τον Καναδά που περιλαμβάνει το, ένα, το νέο σύστημα και η προστασία των επενδύσεων ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει τεθεί σε ισχύ δηλαδή. Πάρα πολύ πρόσφατα ε, επιτύχαμε μια πολιτική συμφωνία επί της αρχής με το Μεξικό, η οποία και πάλι συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά τη νέα ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των επενδύσεων και την επίλυση των διαφορών και ε, μια άλλη συμφωνία που πρόκειται να υπογράψουμε αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι ε, στο παρελθόν ανέκαθεν ε, συζητούσαμε με πολύ διαφορετικό τρόπο την προστασία ε, των επενδύσεων τύπου ναύτα, τύπου TPP, ενώ τώρα ε, εστιάζουμε στην ευρωπαϊκή προσέγγιση και πώς εμείς διαφυλάσσουμε το δικαίωμα αυτό. Βεβαίως είναι ακόμα καθοδόν η διαπραγματεύση με την Ιαπωνία, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί, αλλά εξακολουθούν οι συζητήσεις για την προστασία των επενδύσεων. Βεβαίως έπεται η Ινδονησία, η Χιλή και η Κίνα. Μας είπατε τι έγινε ε, με τις ρήτρε ε, των παλιών κληρονομικών δικαιωμάτων grandfathering. Από το 2015 σας είπα έχουμε μεταρρυθμίσει την προσέγγιση μας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να ε, διαπραγματεύονται και να συνάπτουν διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Θυμίζω ότι τους επιτρέπουμε να το κάνουν αυτό μόνο με εταίρους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαπραγματεύεται προφανώς ή δεν έχει την πρόθεση να το πράξει στο προσεχές μέλλον αυτά όλα δεν θα πρέπει απλώς να είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά να συνάδουν και με την πολιτική μας και την προσέγγισή μας. Γι' αυτό οι πόρους τους επιτρέπουμε να ακολουθήσουν ουσιαστικά την προσέγγιση που έχουμε εμείς στις διμερείς πάντα διαπραγματεύσεις. Επίσης, στην έγκριση πριν τη δώσουμε, περιμένουμε να έχουν ε, μεταρρυθμίσει ουσιαστικά το σκέλος της επίλυσης διαφορών, ε, δεοντολογία, ε, διαφάνεια και ισχυρή ε, αναφορά να γίνεται συμφωνίας ε, στα διαιτητικά δικαστήρια, τα πολυμερία. Από το 2015, 85 νέες διαπραγματεύσεις έχουμε εγκρίνει, 12 έχουν εγκριθεί προς υπογραφή, γιατί χρειάζεται να δώσουμε την άδειά μας δύο φορές στα κράτη-μέλη. Μία για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και μία για να τις τελειώσουν και να υπογράψουν. Αυτό που δεν θέλουμε και δεν περιμένουμε να κάνουν είναι ε, να επαναλαμβάνουν το Διεθνές Σύστημα Διετησίας και Πύλης Διαφορών σε κάθε μία από τις διμερείς αυτές ε, συμφωνίες. Καμιά φορά είναι πάρα πολύ μικρές οι χώρες εταίροι. Αυτό ήθελα να σας πω για τις διμερείς ε, επενδυτικές συμφωνίες. Για τη συνθήκη του ενεργειακού χάρτη που αναφέρατε κι εσείς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια διαδικασία εξχρονισμού τώρα της συμφωνίας αυτής, όπου ενθαρρύνουμε στεναρά τα άλλα μέλη και τη γραμματεία να προχωρήσουν. Εύκολο δεν είναι, ούτε διμερή συμφωνία, είναι πολυμερή συμφωνία. Συμμετέχουν πολλοί εταίροι, συνεργαζόμαστε μαζί τους και προσπαθούμε να προχωρούμε ε, ε, για τον εξχρονισμό αυτό, ιδιαίτερα στους ουσιαστικούς κανόνες για να προχωρήσουμε σε μια ε, σύγχρονη προσέγγιση τη μεταρρυθμισμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπα, δεν θα είναι εύκολο. Αλλά βολιδοσκοπούμε τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις το επόμενο έτος. Οι χώρες αυτές είναι κυρίως χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης για να προχωρήσουν προς τον εξυγχρονισμό του ενεργειακού χάρτη. Και οι περισσότερες ε, διενέξεις και διαφορές προέρχονται από το τμήμα που δεν έχει μεταρρυθμιστεί. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα πολυμερές διαιτητικό δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών και να αφορά και ε, τον ενεργειακό χάρτη. Ο συνάδελφος. Θα και εγώ μερικά λόγια για το πολιτές ε, επενδυτικό δικαστήριο, πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο και κάποια εξωτερικά στοιχεία. Όπως είπατε και εσείς πρόεδρε, η εντολή για τη διαπραγμάτευση εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου από το Συμβούλιο και τη δημοσίευσαν και αμέσω για πρώτη φορά. Έγινε αυτό. Να δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την έγκριση μια απόφαση. Στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου θα τα βρείτε αυτά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ρωτήσατε για τις σχέσεις με τα συστήματα των διμερών επενδυτικών συμφωνιών και διαιτητικών δικαστήριων. τα συστήματα αυτά θα αντικατασταθούν από ένα πολυμερές ε, επενδυτικό δικαστήριο όταν αυτό αρχίσει να λειτουργεί. Ε, ε, συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε και να στείλουμε αυτό το μηχανισμό, αλλά μέχρι να ισχύσει αυτό, ισχύει το παλιό καθεστώς. Όπως λέγει και ο Κάρλος, πρόθεσή μας είναι να αντικατασταθεί το παλιό, τύπου σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους από το νέο και για τα ενεργειακά. Και αυτό ναι, ισχύει και να καλύπτει πάνω από 3.000 διμερείς εμπορικές συμφωνίες. 300 συμφωνίες έχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 700 οι υπόλοιπες. Άρα είναι σύνολο χίλιες. Έχουν ε, αρχίσει οι συζητήσεις για την πολυμερή ε, μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ΠΟΕ, ε, στα αντίστοιχα όργανα, στην ομάδα εργασίας 3. Στις 23 Απριλίου εκείνη την εβδομάδα ήταν η τελευταία συνεδρίαση Πολλές ήταν οι χώρες παρούσες σε αυτή την ομάδα εργασίας, πάνω από 60. Περισσότερες από ότι το Νοέμβριο, δηλαδή είδαμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Επίσης είδαμε ότι πολλά κράτη-μέλη στέλνουν πιο υψηλό βαθμός αξιωματούχους για να συμμετέχουν σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις, άρα τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, σοβαρότερο. Και κάτι άλλο που μπορεί να έχει ε, τη χρησιμότητά του είναι ότι συμμετέχουν εκτός από χώρε και άλλοι ενδιαφερόμενοι. ΜΚΟ ε, και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Τρία είναι τα βήματα. Το πρώτο να δούμε ποιες οι ανησυχίες αν υπάρχουν μετά την επιθυμία ε, να γίνουν μεταρρυθμίσεις και το τρίτο στάδιο είναι η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Στην ομάδα εργασίας τον Απρίλιο ουσιαστικά ολοκληρώσαμε το πρώτο στάδιο, ας πούμε αναλύσαμε τις ανησυχίες και τα προβλήματα και θα ε, φτάσουμε τώρα στη δεύτερη φάση, κατά πόσο είναι επιθυμητές οι μεταρρυθμίσεις, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα τον Οκτώβριο. Για τις ανησυχίες μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές χώρες θεωρούν ότι το παρόν σύστημα χωλαίνει πάρα πολύ. Πολλές χώρες συμμερίζονται την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ισχυρό σύστημα και πολλές χώρες εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη προσφυγής, για την συνέπεια και την προβλεψιμότητα ε, και πολλοί ανησυχούν για ε, την ad hoc φύση του ισχύοντος συστήματος. Λοιπόν, εφόσον ανησυχούμε όλοι τόσο πολύ, καλό είναι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, να βολιδοσκοπήσουμε το κατά πόσο υπάρχει επιθυμία για ε, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά θα συμβούν ε, στην επόμενη συνεδρίαση τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, φέτος. Τελειώνοντας πάρα πολύ σύντομα, επειδή ρωτήσατε κιόλας, για την υπόθεση αχμία και τις ε, διμερείς ε, επενδυτικές ε, σχέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι θέμα εσωτερικής αγοράς. Δεν απασχολεί τη δική μας υπηρεσία. Αλλά στα πλαίσια και υπό το φως της απόφασης ΑΚΜΕΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να τερματιστούν όλες οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ε, εφαρμοστεί και το Σύμφωνο για τον Ενεργειακό Χάρτη. Και δεν ε, θα ισχύσει αυτό το σύστημα επίλυση διαφορών μεταξύ των κρατών μέλων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε εδώ. Υπάρχουν και υποθέσεις ε, κατά της Ισπανίας και υπάρχουν περισσότερα θέματα ενεργειακής χάρτας μεταξύ κρατών μελών και αυτό είναι απαράδεκτο. Μία ερώτηση όμως. Ποια είναι η κρίσιμη μάζα χωρών που χρειάζεστε για το πολυμερές δικαστήριο επενδύσεων. Ήμουνα στο Αμβούργο πρόσφατα, στο οποίο εδρεύει το Διεθνές ε, Θαλάσσιο Δικαστήριο και έχουν τεράστιες αίθουσες και χώρο. Πόσες χώρες χρειάζεστε. Ο Κάρλο ανέφερε το Βιετνάμ, το Μεξικό, τον Καναδά, που έχουμε το σύστημα επίλυσης διαφορών. Υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο ακόμα χρειαζόμαστε λοιπόν. Ευχαριστώ. Καλή ερώτηση και νομίζω ότι είναι κυρίως επιχειρησιακό το ζήτημα. Το τόφλι είναι πόσες χώρες χρειαζόμαστε ώστε να αιτιολογείται η καταβολή μισθών και η σύσταση γραμματείας. Σίγουρα χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς ε, περιμένουμε και τους εταίρους που ανέφερε ο Κάρλος. Ε, αυτοί θα έχουν δεχτεί ε, κατά την άποψή μας το σύστημα αυτό, το επενδυτικό δικαστήριο. Χρειαζόμαστε κάποιους ακόμα για να αιτιολογείται και η, η δημιουργία του. Αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε 100 ή 150 χώρες. Ε, δεν είναι ε, αριθμοί αυτοί που έχουμε στον ΠΟΕ, ας πούμε. Ε, αν μπορέσουμε να έχουμε 40-50 χώρες, θα ήταν καλό. Αυτό θέλουμε. Είναι εντυπωσιακό όμως και πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει ε, στην ομάδα εργασίας για τις μεταρρυθμίσεις. Ε, νομίζω ότι έχουμε τα σωστά ερωτήματα στη σωστή στιγμή. Ευχαριστώ. Ένα, δύο, τρία αιτήματα. Η Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, μετά από τις εξηγήσεις που μου δώσατε, Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι το εσωτερικό σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών μελών δεν είναι αποδεκτό. Επομένως, ο στόχος είναι να ε, αλλάξουν οι εσωτερικές ε, διμερείς συμφωνίες και να μην υπάρχει το σύστημα επίλυσης διαφορών. Αλλά τα κράτη-μέλη σήμερα κάνουν διμερείς συμφωνίες επενδύσεων με σύστημα επίλυσης διαφορών, γιατί ε, το νέο σύστημα θα συστήχιζε πάρα πολύ ακριβά. Και υπάρχει και μία πλαισίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συνοδεύει αυτές τις διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών που γίνονται με τρίτους και εξηγεί γιατί είναι συνεπής με την ευρωπαϊκή πολιτική. Όμως, εάν η ευρωπαϊκή πολιτική θεωρεί ότι το σύστημα επίλυσης διαφορών είναι εκτός παιχνιδιού, νομίζω ότι το αποφασίσαμε αυτό και λέμε ότι το σύστημα επίλυσης διαφορών το ISDS είναι εκτός παιχνιδιού και πώς ε, μπορείτε να θεωρείτε ότι ένα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να, να συνάψει διμερή εξωτερική συμφωνία με σύστημα επίλυσης διαφορών. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της πολιτικής που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την πολιτική που προβλέπετε και πλαισιώνετε εσείς για τα κράτη-μέλη. Τουλάχιστον λοιπόν τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να συνάπτουν διμερή συμφωνίες επενδύσεων με ε, το ISDS. Και φυσικά αυτό έρχεται να προσθεθεί και στην τελευταία απάντηση που ρωτήσατε. Μα αν διευκολύνεται τα κράτη-μέλη και ε, να του πείτε ότι το πολυμερέ δικαστήριο είναι πολύ δαπανηρό, θα μπορείτε να κάνετε σύστημα επιλυση διαφορών. Ε, εάν του απαγορεύσετε να έχουν σύστημα επιλυση διαφορών, θα πάνε πολύ πιο εύκολα προ το πολυμερές δικαστήριο. Αν του πείτε ότι δεν πρέπει να πληρώσετε το ICS ε, και δεν ε, τους απαγορεύσετε να έχουν σύστημα επίλυση διαφορών, δεν θα πάνε ποτέ προ το πολυμερέ δικαστήριο. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη ανησυνέπεια σήμερα για την πολιτική που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη. Είμαι οργισμένη γιατί είμαι από το Βέλγιο που έθεσε και ερώτημα στο δικαστήριο. Ε, υποχρεωτικά πρέπει να, ε, να παραδεχτώ. Αλλά έθεσε ερώτημα όσον αφορά τη συμβατότητα του ICS και η ίδια αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή έχει στα σκαριά, είδα το έγγραφο, ε, μια διμερή συμφωνία με ε, το παλιό σύστημα επίλυση διαφορών. Η ίδια λοιπόν αυτή η χώρα, το Βέλγιο, ετοιμάζεται να κάνει διμερή συμφωνίες με το σύστημα επίλυση διαφορών. Και είναι αλήθεια, αλλά στην πολιτική μπορούμε να είμαστε και υποκριτές, έχουν προσθέσει ένα μικρό κεφάλαιο που λέει «Αλλά εμείς είμαστε υπέρ του πολυμερούς ε, δικαστηρίου επενδύσεων». Ένα, ε, μια φρασούλα έχουν βάλει. Κάνουμε συμφωνία για, με σύστημα επίλυση διαφορών και βάζουμε και μια παραγραφούλα και λέμε ότι εμεί θα προτιμούσαμε το πολυμερέ. Αν θέλετε λοιπόν πραγματικά οι χώρε να πάνε προ το πολυμερέ, υποχρεώστε τι να πάνε προ το πολυμερέ, χωρί να του ε, λέγοντά του ότι δεν υπάρχει καμία συνέπεια αν έχετε ένα σύστημα επίλυση διαφορών, αφού εμεί ω Ευρωπαίοι αποφασίσαμε να το αντικαταστήσουμε με το πολυμερέ δικαστήριο. Η Emma McClarkin. Um, ένα από τα βασικά σημεία του HDS είναι ο ορισμός των ε, ε, διαιτητών στην εμπορική διαιτησία. Πώς θα διορίσετε τα μέλη του Πολυμερούς ε, Επενδυτικού Δικαστηρίου και πώς θα διασφαλίσετε την εξαρτησία τους. Και επίσης θέλω να ρωτήσω πιο ευθέως για μια αφήνεις της κατάσταση στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική, στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα και το Χόγκον και πότε θα το δούμε αυτό να ξεκινάει. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Πρόεδρε, όπως θα γνωρίζετε, δεν είναι υπέρμαχος της προστασίας των επενδύσεων, έτσι όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ξεχωριστό δικαστήριο διαιτητικό για τις επενδύσεις. Αυτό είναι ταξική δικαιοσύνη. Να πηγαίνουν στην κανονική δικαιοσύνη. Ε, και αυτό είναι καλύτερο, πιο αντικειμενικό και πιο δίκαιο από ότι ένα ειδικό διαιτητικό δικαστήριο. Μπορεί τώρα να έχουμε κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με το ISDS για την επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους και το ICS που γνωρίζουμε από το ΣΕΤΑ, αλλά ακόμα δεν ε, έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν ιδιώτες, ΜΚΟ, συνδικάτα, ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ούτε να, ακούσουν, κάνουν τη φωνή τους να γίνει ακουστή. Εν πάση περιπτώσει, μια που το συζητάμε, έχω και κάποιες ερωτήσεις, παρόλο που διαφωνώ. Ο κύριος ε, Μπράουν είπε ότι ενδιαφέρονται πολλές χώρες. Ε, πόσες ενδιαφέρονται και ποιες είναι αυτές. Το ενδιαφέρον είναι <laughs> ένα πράγμα και εγώ ενδιαφέρομαι, αλλά δέσμευση έχει εγώ εκτός από ενδιαφέρον ε, να ασχοληθούν. Και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας, Οκτώβριος, Νοέμβριος μας είπατε. Ε, έχουμε καιρό ακόμα. Από εκεί και πέρα τι. Πότε σκοπεύετε να το ε, στήσετε αυτό το δικαστήριο. Τι γίνεται με τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Συμφωνεί η Ιαπωνία με το ICS. Γιατί υπάρχουν και χώρες που επιλέγουν το σύστημα ε, ΣΕΤΑ. Ε, και τέλος, η Αυστραλία επανειλημμένα έχει πει ότι δέχεται συμφωνία χωρίς καμία τέτοια ρύθμιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το βλέπει αυτό. Ο Κάρλο. Η Δεν ξέρω ποιος. Thank Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις και μετά κάποιες θα τις απαντήσει ο Κάρλο γιατί είναι πιο κατάλληλος. Όσον αφορά αυτό που έθιξε η κυρία Αρένα και θα σχολιάσω και για το Βέλγιο. Δεν θα σχολιάσω το Βέλγιο, μάλλον είναι αρμοδίο του Βέλγιο να αποφασίσει την πολιτική του. Υπάρχουν ε, δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η αδειοδότηση που θα δοθεί από τα κράτη-μέλη είναι για χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διαπραγματευτεί. Αυτό που κάνουμε με τις χώρες που πραγματευόμαστε, αντικαθιστούμε τα BIT των κρατών μελών με πιο εξχρονισμένα υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη όταν διαπραγματεύονται αυτές τις διμερείς ε, συμφωνίες είναι ε, πρέπει να βάλουν υπόψη τις ε, βασικές αλλαγέ, όχι όλες, αλλά κάποιες τις οποίες, ή τις πιέζουμε πρέπει να έχουν έναν κώδικα δεντολογίας, δεν έχουν διαφάνεια να ορίζουν με διαφάνεια τους ε, διαιτητές και να υπάρχει και η, συμφωνία και του άλλου ενδιαφέροντος μέρους. Ε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνοχή αλλά σε επίπεδο και το βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να ζητήσουμε από μικρότερες χώρες να δεχτεί το νέο σύστημα γιατί υπάρχουν και υπάρχει το δυτικό κόστος. Όμως αυτό που έχουμε κατανοήσει είναι ότι πρέπει τα κράτη-μέλη πρέπει να ακολουθούν την ευρωπαϊκή πολιτική και για να υπερσπιστώ το Βέλγιο ήταν πολύ υπεύθυνο στις ζητήσεις και στο Συμβούλιο και στην ομάδα εργασίας για να διασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθεί όντω η σύσταση του Πολυμερούς Επενδυτικού Δικαστηρίου. Είναι μια ιδέα στην οποία, για την οποία έχουμε δεσμευτεί και είμαστε επιπισμένοι ότι θέλουν να το εφαρμόσουν σε όλες τις συμφωνίες και τις υπάρχουσες συνθήκες που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργασιών μας αλλά και τις ε, διαπραγματεύσεις ε, τρέχουσες. Δεν είναι μια ιδανική κατάσταση, όπως είναι μια μεταβατική κατάσταση, όπως προχωράμε προς την δημιουργία ενός ε, πολυμερούς δικαστηρίου επενδύσεων και στην θα γίνει αντικατάσταση των αντιμερών συμφωνιών από αυτό. Σε αφορά την ερώτηση... Ε, κάτι ακόμα. Θέλω να προσθέσει ο Πρόεδρος. Υπάρχει περίπτωση στην οποία δεν επιτρέψατε κράτο μέλος να ξεκινήσει πραγματεύσεις. Ο Κάρλο θα απαντήσει. Συνήθως αυτό συμβαίνει ως εξής. Ε, φροντίζουμε να μην στήσουν ε, άδεια για κάτι για το οποίο δεν θα δώσουμε την έγκριση. Άρα το λύνουμε άτυπα το θέμα μας κάνουν μια άτυπη, μας απευθύνουν άτυπο αίτημα και πολλές φορές τους κάνουμε να αλλάξουν κάποιες διατάξεις ώστε όταν επίσημα υποβάλλουν το αίτημα και επειδή έχουμε και περιορισμένο χρόνο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου δεν έχουν ε, λάβει έγκριση. Um, ε, θα πω ερώτηση της όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού των δικαστών έχουμε κάνει μια διαξυνάμεσα στο επενδυτικό σύστημα και το πολυμερές σύστημα θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της χώρα εταίρου. Έχουμε πέντε ε, Ευρωπαίους, πέντε Καναδούς και πέντε μη Ευρωπαίους συμφώνηση με τον Καναδά να υπάρχουν 15 άτομα. Η Επίτροπος Μάλμστρομ έχει υποσχεθεί στο Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό και τώρα κοιτάμε ακριβώ ποιε θα είναι οι διαδικασίε που θα εφαρμόσουμε για να το πετύχουμε αυτό. Θέλουμε να γίνει μια αυστηρή επιλογή, να υπάρχει διαφάνεια και ότι τα άτομα θα διοριστούν με κατόπιν αποφάσεις του Συμβουλίου μετά από πρόταση της Επιτροπής. Μελετάμε και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά για το πολυμερές δικαστήριο είναι ένα βασικό θέμα. Αυτό υπάρχουν τρία βασικά θέματα. Είναι ένα από τα βασικά θέματα και αυτό, το πώς θα διασφαλίσουμε μια αντικειμενική διαδικασία διορισμού. Θα δώσουμε έμφαση σε αυτό το θέμα, στις διαπραγματεύσεις αν δείτε άλλα διεθνή δικαστήρια, σε δια... στο το ποινικό δικαστήριο, παραδείγματο χάρη, και δείτε πώς διορίζονται τα μέλη, θα δείτε ότι όλα τα σύγχρονα δικαστήρια έχουν ένα screening system όπου οι δεχόμενοι δικαστές εξετάζονται από την επιτροπή που αποτελείται από επιπειραμένους δικαστές και που τους εξετάζουν για να δουν κατά πόσο είναι κατάλληλοι να διοριστούν. Άρα κοιτάμε παρόμοια συστήματα. Αυτό όμω είναι πάλι κάτι το οποίο θα τεθεί από διαπραγμάτευση. Περνώ σε επόμενο ερώτημα για το πόσε χώρε ενδιαφέρονται. Το πλεονέκτημα ε, των ΗΕ, το οποίο στα στην Έθνη, είναι ότι ενδεχόμενα μέλη είναι όλα τα μέλη του ΟΗΕ. Ξέχασα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνείσφερε σε ένα ταμείο ειδικό για να καλύψει τα έξοδα των ταξιδιών από, ε, ανάπτυξη χώρες, πλήρης συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει, ε, υπήρξε μια συνεδρία τον Απρίλιο, είχαμε 60 χώρες, πολλά, πολλές χώρες από την Ελληνική Αμερική και ε, ένα αυξημένο αριθμό αφρικανικών χωρών. Δεν είμαστε σε, στο επίπεδο ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο ώστε να αποφασίσουμε ποια κατεύθυνση θα πάρει η μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ένα δεύτερο βήμα, αλλά σε αυτό θα προχωρήσουμε το Νοέμβριο. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι πολλές χώρες ε, έχουν τις ίδιες ανησυχίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχει δυνατότητα για περισσότερο διάλογο, υπάρχει η πρόθεση να είναι ε, μια δικασία που θα συμπεριλάβει τους πάντες. Το χρονοδιάγραμμα και αυτό το είναι υποσυζήτηση. Δύο φορές το χρόνο θα υπάρξει ε, ομάδα εργασία, δύο φορέ το 2018 και δύο φορέ το 2019. Ε, αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή, να υπάρξουν ε, περισσότερε συναντήσει ε, και να αφήσουμε το τεχνικό έργο για αργότερα. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια. Είναι δύσκολο και θα δεν θα ήμουν ειλικρινής αν ήθελα να σας δώσω μια ακριβή, ένα ακριβή αριθμό. Η Ιαπωνία ναι, είναι πολύ ενεργή στις διαδικασίε, διαδικασίες, στις ε, συζητήσει. Είναι υπέρ της προσέγγισης ε, που θέτησαν στην συμφωνία της, δια, της ε, συμφωνίας για τις δύο πλευρές του Ειρηνικού. Είναι μια πολύ σταθερή στη βαρύ Συμφωνία, αλλά προς το παρόν η θέση τους ε, είναι πιο κοντά στο πρότυπο του TPP. Πολύ ερωτήσει για τον Κάρλο. Το ενδιαφέρον με την Ιαπωνία είναι ότι στο ουσιαστικό κομμάτι ε, καταφέραμε να σημειώσουμε μια καλή πρόοδο, άρα τώρα πιο πολύ θα πρέπει να ασχοληθούμε με ε, το σύστημα διαφορών. για την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Ο αρχικός στόχος ήταν να καλύψουμε την ευρύτερη περιοχή της Κίνας μαζί με και με ένα συμπληρωματικό τρόπο με τη συμφωνία που διαπραγματευόμαστε με την ε, Κίνα η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Βρισκόμαστε ε, στη μέση των διαπραγματεύσεων και είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Hong Kong και την Ταϊβάν είμαστε σε ένα ακόμα πιο πρώιμο στάδιο. Έχουν γίνει συζητήσεις προκαταρκτικές. Ε, ήταν καλές μέχρι στιγμή. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ώστε να κάνουμε κάποια πρόταση αντιπραγματεύσεις. Πρώτα πρέπει να κάνουμε μία αξιολόγηση αντικτύπου και με βάση αυτή να προχωρήσουμε και να το προσφέρουμε στο Συμβούλιο. Σίγουρα η πρόθεση είναι να συμπληρώσουμε την ε, επενδυτική σχέση που θέλουμε να καθιερώσουμε με την ε, Κίνα. Ολοκληρώνουμε και την συζήτησή μας για τις επενδύσεις. Θα παραμείνουμε σε επαφή για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι που παραμείνετε στο τέλος της συνεδρίασης. Θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Καλό απόγευμα.